Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Γιατί υπήρχε πρόβλημα κυκλοφοριακό σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες και φαντάζομαι και άλλοι θα το αντιμετώπισαν. Ευχαριστώ για την υπομονή σας πάντως. Πριν περάσουμε στο πρώτο σημείο της της διάταξης, ο κύριος Κόρπετ θέλει να θέσει διαδικαστικό. Με βάση το άρθρο 162 παράγραφος παράγραφοι 3 και 6 το Κοινοβούλιο αποφάσισε η συζήτηση που θα αρχίσουμε για το Brexit να γίνει μόνο με ένα γύρο μιλητών από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων. Αυτό όμως έχει μια συνέπεια, κυρία Πρόεδρε. Θα ακουστούν τρεις φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία στη συζήτηση. Και όλοι είναι ε, από τους υπέρμαχους του Brexit. Δηλαδή θα ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση ούτε μία βρετανική φωνή από τους πολέμιους του Brexit. Και με, με βάση μάλιστα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ε, η κρατούσα γνώμη πλέον στη βρετανική κοινή γνώμη είναι κατά του Brexit. Κάτι που δεν θα αντικατοπτρίζεται στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόρμπετ. Το σημειώνουμε. Αλλά αυτή ήταν απόφαση των πολιτικών ομάδων να γίνει η συζήτηση με αυτή τη μορφή. Οπότε δεν μπορώ παρά να τηρήσω την απόφαση των πολιτικών ομάδων. Πάντως σημειώνουμε το σημείο που επισημάνατε. Περνάμε τώρα στι δηλώσει Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Υφυπουργό Έτσταντλερ εκ μέρου του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κύριε Επικεφαλή της διαπραγματευτικής ομάδας, κύριε Βαρνιά, κυρίες και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Euratom και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να κάνουν τα απαραίτητα ώστε η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ στι 30 Μαρτίου του 2019. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση ενέκρινε την πολιτική διακήρυξη που θεσπίζει το πλαίσιο για τι μελλοντικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αναφέρθηκε η επιθυμία μας να έχουμε όσο το δυνατό πιο στενή εταιρική σχέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αναφέρεται στη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η έκβαση αυτή θα ήταν αδύνατη χωρίς την δέσμευση, την προσήλωση και την αποφασιστικότητα του κυρίου Μπαρνιέ και του επιτελείου, στον οποίο δώσαμε τα εύσχυμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης υπήρχε μια αίσθηση ενότητας ε, και κοινή ε, ευθύνη από τις 27 χώρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γενικώ μια ενότητα και υπευθυνότητα από όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν επευκαιρία να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έγκαιρη συμμετοχή και τη συνεχή συνεργασία με την ε, κατευθυντήρια ομάδα για τον Brexit και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ε, οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο θα κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει η υπογραφή τις επόμενες εβδομάδες, ώστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη διαδικασία συνένεσης εμπρόθεσμα και πριν το Μάρτιο του 2019. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στον επικεφαλής διαπραγματευτή για τον Brexit, κύριο Μισελ Παρνιέ. Καλώς ήρθατε. Και παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ βεβαίως για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεκινώντας μεταφέρω τις απολογίες του Πρόεδρου Γιουνκέρο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ε, Σύνοδο των G20. Είμαστε σε μια στιγμή κρίσιμη, μια στιγμή μεγάλης σοβαρότητας. Ε, Μερικού μήνε αφού ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσει, των οποίων είχα την τιμή να ηγηθώ υπό την καθοδήγηση και με την εμπιστοσύνη του, του Προέδρου Ζων Κλοντ Ιουνκέρα, αλλά και με την υποστήριξη ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και εσείς κυρία Υπουργέ υπενθυμίσατε, την Κυριακή ε, ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας για την ε, αποχώρηση του Συμβούλιο αλλά και την πολιτική διακήρυξη που προσδιορίζει το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων και θα ήθελα επί τη ευκαιρία και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστώ το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ντόναλτ Τούσκ, ολόκληρη την ομάδα τις ομάδες που ασχολήθηκαν αλλά και τι ε, επακόλουθε προεδρίες με τις οποίες συνεργάστηκα σήμερα την Αυστριακή αλλά και πριν την ε, Βουλγαρική, την Εστονίκη και τη, και τη Μάλτα και θα συνεχίσουμε βέβαια και με τη Ρουμανία στους ε, προσεχείς μήνες. Οι συνομιλίε λοιπόν και οι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία αποχώρηση ε, έχουν ε, ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει αυτό το διάστημα. Έχει έρθει η ώρα πλέον τη κύρωση από την Βουλή των Κοινοτήτων, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη. Πλέον είναι δύσκολε βέβαια οι συνθήκε αυτή τη διαπραγμάτευση και πολύ περίπλοκα όλα τα ζητήματα που εγείρονται με αυτή την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έτσι η συμφωνία αυτή που έχει κατατεθεί, η συμφωνία για τακτή αποχώρηση και πολιτική διακήρυξη είναι η μόνη και η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ένα μεγάλο βήμα το οποίο έγινε δυνατό χάρη στις κοινέ μας προσπάθειες και χάρη σε μια σαφή πολιτική βούλη των 27 κρατών μελών αλλά και όλων των θεσμικών οργάνων. Ιδιαίτερος κυρία Πρόεδρε η συμφωνία Αποχώρηση και η πολιτική διακήρυξη οφείλουν τα μάλα, τα μάλα υπογραμμίζω, στα τέσσερα ψηφίσματα σα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην επαγρύπνηση που επέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή της ε, διαπραγματεύση, από την αρχή των συνομιλιών. Βεβαίω γιατί η προτεραιότητά σα, όπω και η δική μου άλλωστε, ήταν η προστασία των συμφερόντων των πολιτών που εκπροσωπείτε, των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των συμφερόντων τη ενιαία αγορά, αλλά και τη ε, απρόσκοπτης και ορατότητα των τεσσάρων ελευθεριών και της ελευθερία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για δύο έγγραφα τα οποία μαζί χτίσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμφωνία και πολιτική διακήρυξη. Και κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα με, μέσω ημών να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Ταγιάννη και να πω ένα ευχαριστώ προσωπικό στον Κίφερ Χόφστατ, συντονιστή ε, του, εκ μέρους του Κοινοβουλίου για τον Brexit αλλά και σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κυρία Χιούμπνερ, τον κύριο Μπρόκ, τον κύριο Γκουαλτιέρη, την κυρία Ζήμερ τον κύριο Λάμπερτς που εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως μέλη της Επιτροπής ε, ε, παρακολούθησης ε, συνόδεψαν αυτές τις συνομιλίες ε, στο πλαίσιο του Steering Group για το Brexit. Ευχαριστώ πολύ τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, την κυρία Σεσίλια Βίκστρεμ και λέω, εκφράζομαι τι ευχαριστίε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο πέρα ενό δρόμου που είναι ακόμα μακρύ και δύσκολο. Αυτό που προκύπτει ω αποτέλεσμα από την Σύνοδο τη Κυριακή είναι το αποτέλεσμα ταυτόχρονα μια μεθοδική εργασία που από κοινού πάλι οργανώσαμε. Ξεκινήσαμε με τάξη δηλαδή και όπω ήταν λογικό, ξεκινήσαμε από τη Συμφωνία Αποχώρηση, μια τακτή αποχώρηση, πριν αρχίσουμε να συζητούμε το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων με τον Ηνωμένο συμφωνήσαμε προκαταβολικά να διευθετήσουμε ζητήματα τα οποία ήταν και παραμένουν θέματα προτεραιότητα για εσά, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα δικαιώματα των πολιτών, την ειρήνη και σταθερότητα στην Ιρλανδία, το δημοσιονομικό κανονισμό, τη δημοσιονομική διευθέτηση. Και πάνω απ' όλα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εξ αρχή η δουλειά που κάναμε έγινε με απόλυτη διαφάνεια. Άρα σε, απόλυτες, σε συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε. Με τη μέθοδο αυτή λοιπόν μπορέσαμε και να εξηγήσουμε τι ήταν το διακύβευμα σε κάθε περίπτωση, τι ήταν δυνατόν, αλλά και τι δεν ήταν δυνατόν δεδομένων των θεμελιωδών αρχών πάνω στους οποίους στηρίζεται η Ένωση. Εξ αρχής τονίσαμε το πώς πρέπει και μπορούμε να κάνουμε ε, σεβαστές τις αρχές μας πώς μπορούμε και πώς οφείλουμε να κάνουμε σεβαστές τις αρχές μας, αλλά και ποιε, πώς μπορούμε να κάνουμε σεβαστές τις κόκκινες γραμμές που είχε υποδείξει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εν τέλει μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα πεδίο συμφωνίας. Και έτσι, εν τέλει, αυτό το πλαίσιο μπόρεσε να προσφέρει σταθερότητα, ορατότητα, προβλεψιμότητα στις διαπραγματεύσεις αυτές και, αυτές και κανείς δεν μπορεί ε, αντικειμενικά ομιλώντας να εκφράσει έκπληξη ε, για κάτι το αναπάντεχο που προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις. Ξεκινώντας βεβαίω θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επεθύμησε τον Brexit. Άλλωστε κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει μπορέσει να επιδείξει θέμενη αξία του Brexit. Αλλά σεβόμεθα τον, ε, την δημοκρατική και κυρίαρχη επιλογή του Βρετανικού λαού και όπως και η Βρετανική κυβέρνηση ζήτησε ετέθησε και κίνηση αυτή η διαδικασία για μια τακτή οργανωμένη αποχώρηση. Πάντως τα δύο έγγραφα της Κυριακής επιτρέπουν τον περιορισμό των ανετικών συνεπειών του Brexit και για τις δύο πλευρές και ιδιαίτερο και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συμφωνία Αποχώρησης εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για κάθε ε, φυσικό και νομικό πρόσωπο και για τις περιφέρειες ε, που ε, θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες από την αποφάση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση, ιδιαίτερα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4,5 εκατομμύρια που διαμένουν στο, Ευρωπαϊκό, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα τους κατοίκους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Και επίσης ε, κάθε διάσταση ανθρώπινη, κοινωνική, οικονομική της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένου Βασιλείου Βορρά Νότου δεν θα λησμονηθεί. Το backstop στο οποίο έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή η αποφυγή της επαναφοράς μιας της επαναφοράς των συνόρων, των υλικών συνόρων, των σκληρών σύνορων στην ε, Βόρεια Ιρλανδία ε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική λύση. Επίσης, πολλά είναι τα έργα από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και τόσους άλλους που αναλαμβάνονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαστήρια, πανεπιστήμια ε, που εποφελούνται. Όπως και οι γεωργοί εποφελούνται από την κοινή γεωργική πολιτική και ήθελαν και αυτοί να εξασφαλιστεί η να, να προστατευτούν τα δικαιώματά του σε βιομηχανική ιδιοκτησία πέραν τη γεωργραφικής προέλευση. Όλα αυτά μαζί με τι επιχειρήσει που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τομεί ε, για μα, ε, ξεκινώντα βέβαια από, τα, από τους πολίτες, από τα άτομα στου οποίου πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκε βεβαιότητα, εκεί που το Brexit προξενεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Και έτσι λοιπόν αυτή η πολύ πυκνή τόντη το παραδέχομαι συμφωνία αποχώρησης γιατί πρόκειται για μια νομική πολύ επακριβή και περίπλοκη ε, συμφωνία ε, σε αυτό ακριβώς στοχεύει. Η δεν νομική, ε, η πολιτική διακήρυξη ορίζει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για τις περαιτέρω σχέσεις. Διαπραγματεύσεις μέσω των οποίων σας διαβεβαιώ κύριε και κύριοι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υπεραμείνεται των δικαιωμάτων, των συμφερόντων της και να στηρίζει τις ίδιες αρχές. Οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διαπραγματευτής σας θα υιοθετήσουν την ίδια στάση που είχαμε μέχρι τώρα, επιθετικότητα δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν θα υπάρξει ποτέ. Εκδικητικότητα δεν υπήρξε ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Δεν υπήρξε όπως και δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει πνεύμα ε, τιμωρητικό ε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένο Βασίλειο, να αγωνιζόμαστε μαζί του για να χτίσουμε αυτή τη μελλοντική σχέση και να χτίσουμε αυτή τη ε, συμφωνία μέσα σε πνεύμα σεβασμού, όπω τον οφείλουμε σε μια χώρα μεγάλη που πιστεύουμε ότι θα πρέπει θα μείνει και εταίρο και φίλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις μελλοντικέ αυτές σχέσεις λοιπόν και οπωσδήποτε δεδομένου ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αποχώρηση του Ενωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενή αγορά, προφανώς δεν μπορεί να παραμείνει το status quo ante. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι επιχειρήσεις και να προετοιμαστούν αναλόγω. Κοινή μας βούληση πάντως είναι να χτίσουμε μια εταιρική σχέση φιλόδοξη για τι εταιρείε, τις υπηρεσίες, την ψηφιακή οικονομία, την κινητικότητα, τις μεταφορές, τις δημόσιες ε, προμήθειες, την ενέργεια, την εσωτερική ασφάλεια και βεβαίως για τη σταθερότητα στην Ήπειρό μα, την εξωτερική πολιτική. Με μια χώρα η οποία παραμένει δραστηρία οπωσδήποτε και στο Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και στην άμυνα πάνω από όλα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Όσο πιο, καλές, όσο πιο προχωρούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, τόσο πιο πολύ θα είναι ε, και η επαγρύπνησή μας για την εξασφάλιση ενός ότιμου πεδίου αν λοιπόν μπορέσουμε, και επιτρέψτε μου εδώ να πω, ότι όταν μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε, αν μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την πολιτική αυτή διακήρυξη όλες τις διαστάσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η εταιρική σχέση που θα χτιστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια εταιρική σχέση άνευ προηγουμένου και ως προς την έκταση και ως προς το φάσμα τομέων που θα καλύπτει. Όπως θέλησε και ο πρόεδρος Γιονκέρ, τα κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προετοιμαζόμεθα. Και θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον αρκτήριο λάκτισμα για αυτή την ε, διαπραγμάτευση άπαξ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετατραπεί σε τρίτο κράτο, σε τρίτη χώρα. Βεβαίω, κυρία Πρόεδρε, παραμένει ένα στάδιο καθοριστικής σημασίας η κύρωση της συμφωνίας αποχωρηση Έχει έρθει πλέον η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνε του. Οι βουλευτέ του Ηνωμένου Βασιλείου θα κληθούν τις επόμενες ημέρε να τοποθετηθούν για τη συμφωνία αποχώρηση και την πολιτική διακήρυξη. Ψήφος δε, η οποία δεσμεύει τη χώρα τους για το μέλλον. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε, εγώ θα σεβαστώ τον, ε, τη συζήτηση, τον χρόνο για τον πολιτικό διάλογο, την πολιτική συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Κοινοβούλιο, αλλά βεβαίω ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και η κύρωση, πρέπει να δοθεί και ο χρόνο για την κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμμετέσχει και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο τη διαπραγμάτευση και που τελικά εσεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχετε την τελευταία λέξη. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Βαρνιέ. Και τώρα να περάσουμε στους ομιλητές ε, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο συντονιστής για θέματα του Brexit, ο κύριος θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω και να χαιρετήσω τη συμφωνία αποχώρησης ως πολιτική δήλωση. Νομίζω ότι μπορούμε εύκολα σήμερα να δηλώσουμε ότι και οι δύο βασίστηκαν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς οι τέσσερις ελευθερίες οι οποίες υποστηρίζουν την ενιαία αγορά και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζει με αυτόνομο τρόπο. Είναι σημαντικό όμω να διευκρινιστεί στη συζήτηση αυτή ότι υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία τα οποία λήφθησαν υπόψη. Το πρώτο είναι ασφαλώ οι θέσει, οι κόκκινε γραμμέ ενδεχομένω του Ηνωμένου Βασιλείου και τη κυβέρνησή του μετά την απόφαση να τερματιστεί η συμμετοχή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει τη συμφωνία αυτή τις συμφωνίες αυτές μάλλον κάτι συχνά το παρά που το προβλέπουμε είναι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συμφωνία του 1998, η συμφωνία αυτή κατέστη ε, δυνατή μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό καταδεικνύει, θεωρώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς είναι ε, και σημαίνει πάει επανασυμφιλίωση, τέλος της βίας, ειρήνη. Τα αποτελέσματα όλων αυτών αποτυπώνονται στην ε, συμφωνία τη αποχώρηση. Θεωρώ ότι είναι τη βέλτιστη συμφωνία, λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία μόλις σα περιέγραψα. Και για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, ε, μάλλον για την επιτυχία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ για την πρώτη φορά τον Μισελ Μπαρνιέ. Προσωπικά έκανε τεράστιο ε, έργο σε στενή συνεργασία με το Κοινοβουλίο και με την ε, σχετική ομάδα και θα ήθελα να συγχαρώ και όλα τα μέλη της ομάδα τη Επιτροπή για το Brexit, πέρα από τι γραμμέ των πολιτικών κομμάτων, θεωρώ ότι η δουλειά ήταν πάρα πολύ καλή που έγινε. Τα αποτελέσματα λοιπόν τώρα. Το αποτέλεσμα, Μισελ, είναι τριπλό ε, ω προ τα αποτελέσματά του. Καταρχά, να περιορίσουμε στο βαθμό του δυνατό τι στρεβλώσει ε, και για τι δύο πλευρέ, κυρίω σε ό,τι αφορά την οικονομία. Να υπάρξει μια τακτή λοιπόν αποχώρηση και ένα χρονικό περιθώριο 2 έω 4 ετών για να ολοκληρωθούν Ήδη διαπραγματεύσει για τι μελλοντικέ σχέσει. Δεύτερο αποτέλεσμα, να αποφύγουμε σκληρά συσσαγωγικά σύνορα με την Ιρλανδία και να διατηρηθεί η ειρήνη και τα όσα μένουν από την ε, Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και ήταν μεγάλη μας προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρηθούν τα δικαιώματα όλων μας των πολιτών. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια και την υποστήριξη των διαπραγματευτών μας, θεωρώ ότι βελτίωσε σημαντικά την ε, πρόταση και τη συμφωνία. Και πέραν τούτου, είμαστε δεσμευμένοι Πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία συνένεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λάβαμε από, να λάβουμε από τους Βρετανούς α, ε, ομολόγους μας ε, διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα πιστεύω ότι η συμφωνία αποχώρησης και η πολιτική διακήρυξη μας δίνει την ευκαιρία στο μέλλον να διαμορφώσουμε στενές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Η βάση λοιπόν όπως είπατε και στη συμφωνία και στην πολιτική διακήρυξη, είναι μια συμφωνία εταιρική σχέση, σύνδεση. Αυτό είχε προτείνει άλλωστε από την πρώτη μέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν μια τέτοια συμφωνία, σύνδεση, συμφώνησε και η Βρετανική κυβέρνηση. Γιατί θα εφαρμοστεί με προσωρινό τρόπο όταν θα σε εφαρμογή μετά την εφαρμογή και την έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επικυρωθεί σε έναν γύρο επικύρωσης από τα κρατημέλη μελη προκειμένου να αποφευθούν οι περιπλοκές της σχέσης μας, για παράδειγμα, με την Ελβετία, που δεν βασίζεται σε μία συμφωνία σύνδεσης εταιρικής σχέσης, αλλά σε ένα συνοθήλευμα συμφωνιών. Η ομάδα, λοιπόν, καθοδήγησης για το Brexit, μαζί με όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσει να εξετάζει την συμφωνία αποχώρησης και την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση ως τμήμα της ε, συμφωνίας, της διαδικασίας ε, συνένεσης και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κοινή επιτροπή. Αυτή η κοινή επιτροπή, κύριε Φερχόφστατ, ε, λέει η Πρόεδρος, είμαι η Πρόεδρος και εγώ θα καθορίσω τα χρονικά όρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθοδήγησή σα, αλλά παρακαλώ να γίνει σεβαστή η Προεδρία. Ναι, και κλείνω άλλωστε Πρόεδρε, λέει ο κ. Φερχόφστατ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα εξετάσει την ε, λειτουργία της κοινή Επιτροπής. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσει που θα λάβει αυτή η κοινή Επιτροπή είναι νόμιμέ. Και όπου αυτό ε, χρειάζεται θα ζητούν και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να έχουμε μια σχετική συμφωνία με το Συμβούλιο. Κλείνοντα να πω ότι δεν υπάρχουν ε, νίκητε, θεωρώ ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια αποτυχία για όλου, και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, η προηγούμενη Κυριακή ήταν μια ημέρα λύπη για όλου. Α ελπίσουμε ότι στο μέλλον ε, η μελλοντική γενιά στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει να ξαναμπεί στου κόλπους τη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βερχόφσα. Το κύριο Μπρόκ. Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου και συνάδελφοι, το Brexit είναι ευρωπαϊκή υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μεγάλο ζήτημα. Πιο πολύ για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, αλλά και για μα είναι μεγάλη υπόθεση. Και γι' αυτό λοιπόν η Κυριακή, όπως είπε ο Γκί Φερχόφστατ, που τον ευχαριστώ για την συνεργασία, σωστά είπε λοιπόν ότι ήταν μέρα λύπηση η Κυριακή. Αλλά βάσει τη διαπραγματευτική ικανότητα του Μισελ Μπαρνιέ και τη ομάδα του, χάρη στην υπομονή του, χάρη στην ε, ικανότητά του, καταφέραμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά τη συμφωνία και να πούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διχασμένο, η κυβέρνηση και ολόκληρη η χώρα. Συμφώνησε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 χώρε. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή συμφώνησαν και απόδειξαν, απέδειξαν ότι είμαστε ενωμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι η ζημία αυτή για την Αγγλία κατέστησε σαφές και με τις δηλώσει της Εθνικής Τράπεζα χθε. Πρόκειται να ακολουθήσει μεγάλη απώλεια ε, στην ανάπτυξη λόγω του Brexit. Αυτή ήταν η χθεσινή δήλωση της Bank of England. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να λέει ότι ψέματα θέλει στη χώρα του. Αυτό δεν αλλάζει όμως τα γεγονότα και διαπιστώνουμε ότι αυτό σημαίνει και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι υποστηρίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις Ή αυτή η συμφωνία ή καμία συμφωνία. Δεν θα ξεκινήσουμε να την απορρίπτουμε, να ξανακάνουμε διαπραγματεύσει και αυτού ξανά από Όχι, αυτή είναι η συμφωνία. Από εκείνη τη διαπραγματευτήκαμε και θα πρέπει να είναι σαφές ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι η βάση για μια μεταβατική φάση. Γιατί έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά αυτό δεν είναι σαφές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης δεν θα υπάρξουν μεταβατικές ε, ε, διατάξεις. Θα είναι ξαφνική και απότομη η αποκόλληση. Με τη συμφωνία λοιπόν ε, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι Πρόκειται για μια δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση για όσους είναι υπέρ της ε, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν απορρίψουν λοιπόν τη συμφωνία αυτή και ενδεχομένως ζητήσουν δημοψήφισμα, είναι πολύ επικίνδυνο και θα απέθυνα έκκληση και προς τις δύο πλευρές λοιπόν να εγκρίνουν αυτή την ε, συμφωνία. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με τα δικαιώματα των πολιτών που θα πρέπει να διατηρηθούν σε ό,τι αφορά την ε, προγραμματισμό ζωής που έχουν, ότι δεν θα υπάρξουν σκληρά σύνορα με τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε αυτό στην οικονομία και στη ζωή των ανθρώπων στην Ισλανδία και στην Βορειολανδία. Και σκοπός του backstop είναι να μην τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό θυμίζω ότι είναι ε, γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρξει κατάχρηση του μέτρου αυτού ούτε στη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρώ ότι οι μελλοντικέ ε, σχέσεις είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να δείξουμε ε, πραγματικά ευαισθησία για μια κοινή λύση δεν θέλει να είναι μέλος της ενιαίας αγοράς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν θέλει τόσες ε, μεγάλες ε, ελευθερίες. Αλλά θέλει να συμμετέχει και η Τερίζα έχει δίκιο. Λέει ότι όσο πιο, πιο παρόμοια πρότυπα έχουμε, τόσο πιο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στις αγορές ο Και γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές θα πρέπει να φροντίσουμε ότι αυτή η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να ευτερηθεί σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να είμαστε σε ίσο επίπεδο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να έχουμε μια κοινή πολιτική άμυνας και προστασίας. Αυτό το θέλουν και οι δύο πλευρές και γι' αυτό λοιπόν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τους ε, όρους πλαίσιο για να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των λαών μας και αυτό ισχύει και για την έρευνα, η κατάσταση των Βρετανικών πανεπιστημίων, των ερευνητικών προγραμμάτων στον Ηνωμένο Βασίλειο. Τελευταία παρατήρηση κυρίε και κύριοι. Ο κύριος Τραμπ χθε βγήκε και δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει ε, σε αυτή τη συμφωνία αποχώρησης. Ο κύριος Τραμπ θέλει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να απομονωθούν, να διχαστούν, προκειμένου να κάνει αυτός ό,τι θέλει από εκεί και πέρα και να τις διχάσει. Αυτά που είπε ο Τραμπ είναι ο καλύτερος λόγος και η καλύτερη εξήγηση για το τι, για το λόγο που χρειαζόμαστε στο μέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να προσπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην αφήσουμε να μας καταστρέψει ο κύριος Τραμπ. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Μισελ, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, η Συμφωνία της Κυριακής θέτει τις βάσεις για μια έφτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε έτοιμοι να κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ Μπαρνιέ για την καταπληκτική του προσπάθεια, για το καταπληκτικό πολύ αξιόλογο έργο του ίδιου και το επιτελείο του σε αυτή την ιστορική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε. Βέβαια δεν μπορώ να κρύψω τη βαθύτατη θλίψη μου για την επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα μα σέβεται την απόφαση αυτή, αλλά εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη τη. γιατί θεωρούμε ότι είναι ιστορικό σφάλμα αυτή η απόφαση και στα μάτια μα θα είναι μια κατάσταση που όλοι θα βγούμε χαμένοι. Και παρά την απογοήτευση και τη ματέωση που νιώθουμε, ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι από την αρχή ε, αναλάβαμε τις ευθύνες μας και δείξαμε υπευθυνότητα και σεβασμό και εργαστήκαμε καταπώνητα για πάνω από μία διετία για να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν ε, επηρεαστεί περισσότερο από την απόφαση και να μετριάσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Και αυτό επιτεύχθη χάρη στην καθοδήγηση των, ε, της διαπραγματευτικής ομάδας και χάρη στην ενότητα ε, των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γκίφερ Χόφστετ και όλα τα μέλη της, ομάδα, της διευθύνουσας ομάδας για τον Brexit και ήμασταν πάντα ενωμένοι. Ήμασταν υπεύθυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντα τα θεμέλια για μια έφτακτη αποχώρηση, χωρί καμία αίσθηση εκδίκηση ε, ή καμία απέχθεια. Αλλά ε, θα ήταν ε, ε, έλλειψη σεβασμού απέναντι στου πολίτε να μην εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το συμφέρον τη. Και αυτή η αίσθηση τη υπευθυνότητα θα μα κατευθύνει και στο μέλλον. Θα πρέπει όμω να αποσαφηνίσουμε το εξή. Εναλλακτική λύση σε αυτή που συμφωνήθηκε την Κυριακή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική συμφωνία. Η λήψη υπόψη των κόκκινων γραμμών των Ηνωμένων Βασιλείου μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η μόνη δυνατή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών, την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και της Θελωνιακής Ένωση και αποτρέπει ένα σκληρό σύνορο στο, στην ίσο της Ιρλανδίας με σεβασμό όλων των τμήματων της Συμφωνίας τη Μεγάλης Παρασκευής. Τα δικαιώματα των πολιτών ήταν από την αρχή ύψιστη προτεραιότητα μα και βέβαια το έργο μα εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ε, επαγρυπνούμε για να σεβαστεί αυτό το τμήμα της συμφωνίας, για να γίνει σεβαστό αυτό το τμήμα της συμφωνίας. Ε, ε, και θα ήταν κρίμα να πέσουμε ε, θύματα μιας ε, κακής πολιτικής. Η πολιτική διακήρυξη που συνοδεύει τη Συμφωνία Αποχώρησης αποτελεί το πλαίσιο και τη βάση για μια φιλόδοξη, ευρεία και εμβριθή εταιρική σχέση που θα πάρει τη μορφή μια συμφωνία σύνδεσης και που θα σέβεται πλήρως την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και την αυτονομία της ένομης μας τάξης. Και φυσικά θα έχουμε και ε, τις ε, ερμηνευτικές ε, διακηρύξεις του Συμβουλίου που θα ε, θεωρηθούν νομικά δεσμευτικές και για το Γιβραλτάρ. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές σχέσεις, διευκρινίσαμε τις κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών και τις σεβαστήκαμε και στη διαπραγμάτευση δείξαμε μεγάλο βαθμό ελαστικότητας και κάναμε όσο πιο ελαστική γίνεται τη συμφωνία για να λάβουμε υπόψη τη θέση και του περιορισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε πει ανέκαθε και το επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάξει γνώμη, οι αγκάλε μα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτέ στο μέτρο όμως που θέλετε, να αποχωρήσετε από την ενιαία αγορά και να μην εφαρμόζετε τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων, αυτή είναι η μόνη δυνατή λύση, αυτό είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να φύγετε εφτάκτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας σοβαρή, ε, τη σοβαρή διατάραξη ενός ε, σενάριου χωρίς συμφωνία. Και θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα όρια χωρίς ε, να διακυβευθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προσιλωμένο στις σχέσεις ε, ε, και τους δεσμούς με τις χώρες και τους λαούς μας και γι' αυτό θα παίξουμε προορατικό και δραστήριο ρόλο για να διασφαλίσουμε την ακυριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσουμε θετικές μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ κύριε Γουαλτιέρο, Βανόρντεν. Χωρίς μικρόφωνο. Είναι πολύ εμπειρογνώμονος εδώ για την ιστορική πολιτική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε ότι το Brexit δεν αφορούσε μόνο την οικονομία. Αφορούσε πολύ περισσότερα πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα σε πολλούς άλλους τομείς ε, και τον, ε, έχει παρέμβει όπως ιδιαίτερα ε, εσωτερικά θέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και επειδή ο Βρετανικό λαό ήταν όλο και πιο δυσαρεστημένο με την υπόθεση αυτή, ψήφισε τον Brexit. Λέτε, δεν θέλατε τον Brexit, αλλά δεν κάνετε και τίποτα για να το αντιμετωπίσετε. Ωστόσο, πρέπει να σα πω εγώ. Ε, θα υπάρξουν συνέπειες λοιπόν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο στη Βρετανία. Φαίνεται ότι εδώ ασχολούμαστε πολύ με το να κάνουμε προβλέψεις για τις συνέπειες στο Λονδίνο και τις συνέπειες ε, του Brexit ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ήταν καλό να κοιτάξουμε τι συνέπειες θα φέρει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μια κακή συμφωνία ή κακές μελλοντικέ σχέσεις. Βεβαίως η Βρετανική κυβέρνηση κυβερνηση ερχεται τι διαπραγματευσει σε πνεύμα καλό συνεργατικό, προσβλέποντας σε μελλοντική εταιρική σχέση και έχουμε εξαφνιαστεί στο Λονδίνο από την νομικίστικη και δικολαβίστικη προσέγγιση που επεκράτησε τελικά. Ξέρουμε όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί όποτε θέλει να κάμψει και να, και να παραγνωρίσει τους κανόνες τη όποτε τη βολεύει. Φαίνεται ότι ορισμένες χώρες έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν μια στενή και ιδεολογικά φορτισμένη προσέγγιση υπερασπιζόμενες το ε, εγχείρημα, της, το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως όλο και περισσότερο απορρίπτουν οι πολίτες στον κόσμο και κάποιες από τις μεγαλύτερες χώρες μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητά κατα, ε, κατακρίνουν. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να δίνεται σαν απάντηση στο Brexit ότι πρέπει να προχωρήσετε σε, σε περισσότερη Ευρώπη και πρέπει να σας πω ότι πολλοί είναι αυτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατεπλάγησαν και αισθάνθηκαν και προσβολή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και την αλαζονία. Έτσι λοιπόν, ε, με μια παράξενη, παράδοξη αλληλουχία ε, διαδικασιών που επιβάλλατε, χάσαμε δύο χρόνια. Χάσατε δύο χρόνια, όλα τα άλλα θα είχαν μπορέσει να ολοκληρωθούν. Δεν χρειαζόταν να γίνουν όπως τα κάνατε εσείς. Και έτσι είναι πολύ πιο απαραίτητο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε ταχύτερα σε διαπραγματεύσει για τη μελλοντική σχέση για να καταλήξουμε σε σύντομες, σύντομα σε συμφωνίε, αλλά χρειάζεται και ευελιξία ταυτόχρονα, εγγυήσει δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ε, και τα μελήματα που έχουν διατυπωθεί. Χρειάζεται να αναπτυχθεί ε, ατμόσφαιρα εμπιστοσύνη και καλή βούληση από πλευρά σα, εάν πρόκειται να έχουμε αυτή την καλή σταθερή ε, μελλοντική σχέση που φαίνεται πω τουλάχιστον ε, που από ό,τι φαίνεται όλοι οι πολίτε απαιτούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάμπερτ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε οι συνάδελφοι, οι, πολυ... οι συνάδελφοι με ρώτησαν αν αισθάνθηκα λύπη την προηγούμενη Κυριακή στο Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι αισθάνθηκα ευγνωμοσύνη προ τον Μισελ Μπαρνιέ και την εξαιρετική του ομάδα. Όχι μόνο δηλαδή διαπραγματεύτηκαν την ε, συμφωνία έχοντα υπόψη και γνώμονα το κοινό συμφέρον χωρί ποτέ να χάσουν το θάρρο και την αποφασιστικότητά του, αλλά ταυτόχρονα οργάνωσαν αυτήν την διαδικασία σε ισότιμη, με ισότιμη αντιμετώπιση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω, η συμφωνία δεν είναι τέλεια όπω ε, το βλέπουμε Εμεί, οι πράσινοι θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε ε, πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα και όχι κίνδυνο για οπισθοδρόμηση ως προ τα κοινωνικά ζητήματα, η Τελωνιακή Ένωση κτλ. Και θα θέλαμε πιο ε, οδηγίε για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε αυτό να μην μετατραπεί σε ένα φορολογικό παράδεισο ή μια χώρα νομοποίηση παράνομων εσόδων. Και σα διαβεβαιώ ότι εμεί θα επαγρυπνήσουμε και στο μέλλον γι' αυτό. 18 μήνε λοιπόν πολύ σκληρή δουλειά για να βρεθεί μια συμφωνία. Εάν αυτό δεν είχε καταστεί δυνατό, η χειρότερη εκδοχή που θα ήταν να φύγει με μια ε, παταγώδη έξοδο χωρί να υπάρχει συμφωνία του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καταστροφή για όλου. Χωρί συμβιβασμού λοιπόν για την ακεραιότητά τη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και χωρί. Ε, ε, και με ρεαλισμό από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου συνήφθη αυτή η συμφωνία και αυτό μα φέρει μια κάποια ανακούφιση. Βέβαια, πρέπει να δούμε αν η Πρωθυπουργό θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία για την κύρωση τη ομάδα σε επίπεδο Βουλή των Κοινοτήτων. Για του υποστηρικτέ του Brexit, θα πω το εξή: Εάν το Brexit είναι αυτό που θέλατε και αν παρόλα αυτά θα θέλατε να διατηρήσετε τη συμμετοχή τη χώρα στην ενιαία αγορά, άλλη λύση δεν υπάρχει για εσά. Συμφωνία δεν υπάρχει. Όποιο και να έρθει να διαπραγματευτεί, να αναλάβει τη διαπραγμάτευση εκ μέρου του Ηνωμένου Βασιλείου, θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα ίδια όρια, με του ίδιου περιορισμού που αντιμετώπισε και η Τερέζα Μέη και νομίζω ότι κανεί δεν θεωρεί ότι είναι καλύτερο να αποχωρήσει τον Ηνωμένο Βασίλειο χωρί συμφωνία, γιατί αν το έπρεπε αυτό θα παραβίαζε και τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Ταυτόχρονα δηλαδή επανέ, θα επανέφερε σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία, στην ίσο τη Ιρλανδία και ταυτόχρονα θα παραβίαζε και τι δημοσιονομικέ δεσμεύσει που έχει αναλάβει υπό τι ε, συνθήκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προκύπτουν από την ε, περίοδο κατά την οποία είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορείτε με ό,τι αποχώρηση και να επιλέξετε να απαλλαγείτε των ε, οικονομικών σας υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν ε, Brexit χωρί συμφωνία ε, θα σήμαινε μηδέν ιστοπηλίκων. Άρα η μόνη λύση είναι Brexit με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί τώρα ή Brexit Νιέτ, Brexit χωρίς Brexit δηλαδή. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι φαίνεται πως τα το, το κύριο κόμμα στον Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι διχασμένο στην υπόθεση αυτή. Γι' αυτό καλό ήταν να βρείτε μια λύση. Ε, βρίσκεστε σε πολύ δυσκολότερη θέση εσείς που υποστήριξε τον Brexit. Το Ηνωμένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την εθνική κυριαρχία και αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα και ε, πάτημα στον κόσμο, στο διεθνές σκηνικό, πρέπει όλοι να δούμε μαζί. Ε, θα υπάρξει άλλη πλειοψηφία, δεν ξέρω, μπορούμε να τους ρωτήσουμε, δεν ξέρω. Πάντως, αν υπάρξει δυνατότητα για διαφορετικές πλειοψηφίες, θα είναι πολύ περιορισμένε αυτές τις δυνατότητες. Και είμαι βέβαιο ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να παρετηθεί τις ε, δυνατότητες, τις δυνατότητας του για αποχώρηση, επιλογής του για αποχώρηση, θα είναι ευπρόσδεκτο να παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνοντα Πρόεδρε, θα ήταν απολύτω ανεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλήξει να βγει χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παταγωδός όπως λέω είτε επειδή το θέλησε είτε ε, άθελά του. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Το Συμβούλιο στην ε, συνεδρίαση του στο Συμβούλιο την προηγούμενη Σαββατοκύριακο υπέγραψε τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, στην παρούσα φάση, κανεί δεν μπορεί να πει κατά πόσον με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο πιθανό ένα τακτικό Brexit. Είναι σημαντικό από πλευρά των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστούμε στο χειρότερο σενάριο. Μια κατάσταση που δεν θα υπάρξει συμφωνία. No deal σενάριο. Για την ε, ομάδα καθοδήγηση για τον Brexit και σε ό,τι αφορά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του προηγούμενου έτους δεν ήταν τα πράγματα αυτά ξεκάθαρα και αυτονόητα. Η απόφαση να υποστηρίξουμε αυτή την πλατφόρμα και να συμμετάσχουμε ως, link, ως αριστερή παράταξη στην ε, ομάδα αυτή του Κοινοβουλίου ήταν σωστή. Και θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία με τον Μισελ Μπαρνιέ έθεσε πρότυπα σε ό,τι αφορά τη μελλοντική συνεργασία με τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ήδη τώρα είναι ότι η συμφωνία αποχώρησης δεν είναι κάτι για να γιορτάσουμε. Ανησυχούμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Θεωρούμε ότι τα δικαιώματα δεν είναι τόσο κατοχυρωμένα που να παρέχουν πραγματικά νομική βεβαιότητα για όσου ενδεχομένω θα πλεχθούν από το Brexit. Αυτό που δεν είναι στεγανό στη συμφωνία αποχώρησης δεν μπορεί φυσικά να, να διευκρινιστεί και να διασφαλιστεί με προθέσεις ε, ε, με δηλώσεις προθέσεων. Γιατί στη συμφωνία ε, συμφωνήθηκε και το backstop και έτσι αποφεύθηκε το σενάριο τρόμου στην ε, Ιρλανδία. Το backstop δεν πετυχαίνει αυτό που μας είχαμε υποσχεθεί στην κοινή έκθεση του προηγούμενου Δεκεμβρίου. Το σύνορο μεταξύ με την Ιρλανδία θα είναι πιο σκληρό. Θα διακυβευθούν τα δικαιώματα τα οποία μα είχαμε εγγυηθεί στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Όπως ε, και την Τερέζα Μέη μας απασχολούν ε, οι φωνές αυτών που αμφιβάλλουν και αμφισβητούν τους ε, εξασφαλίζει ότι θα σταματήσει η μεταφορά μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς ε, όμως δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αλλά και ακόμα οι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ ότι υπάρχει ο όρος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ξεχνούν όλοι αυτοί ότι αφαιρούν δικαιώματα και από τους πολίτες τους δικούς τους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που και μετά το Brexit θέλουν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να ζήσουν, θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους πολίτες του υπόλοιπου κόσμου. Μετά την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το είπαν πολύ σήμερα αυτό, θέλουμε να έχουμε στενές ε, σχέσεις. Αυτό το υποστηρίζουμε, αλλά για να μην μείνουμε στα κενά λόγια θα πρέπει να πέσει σκληρή δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με τον Κίφερ Χόφστατ προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για τα δικαιώματα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση έναντι των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να το πω ξεκάθαρα αυτό και θα συνεχίσουμε να το τονίζουμε και στο μέλλον όπως και το θέμα της Βορείου Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάρας έχει το λόγο. Δεν αμφιβάλλω ότι αυτή η συμφωνία αποχώρηση είναι καλή συμφωνία. Είναι καλή συμφωνία γιατί περιέχει μεγάλη μεταφορά χρημάτων. Γιατί διατηρεί την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Γιατί κρατάει την Ευρωπαϊκή, την ε, στην Ελληνική Ένωση και κυρίω το βασικό σημείο, όπω είπε σήμερα το πρωί ο κύριο Μπαρνιέ, υπάρχει και αυτό το backstop, το οποίο σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να το κρατήσουν όμοιρο για πολλά χρόνια. Είναι καλή η συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Ενωμένο Βασίλειο νομίζω ότι είναι η πιο κακή συμφωνία στην ιστορία μα. Κάτι το οποίο ο κύριος, ε, κύριε Μπρόκ το σημείωσε ο κύριο Τραμπ αλλά ξέρετε ότι σέβεται ιδιαίτερο τα μεγάλα εθνικά κράτη της Ευρώπης και δεν είναι εχθρός κανενός από αυτά. Κύριε Μπαρνιέ, μακάρι να είστε στα δική μας πλευρά, γιατί ε, παίξατε το παιχνίδι και δεν πιστεύετε την τύχη σας ότι βρεθήκατε αντιμέτωπος με τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό και πετύχατε όλα όσα θέλετε και εξαπατήσατε το βρετανικό κοινό και Συμφωνήθηκαν όλα αυτά σε 38 λεπτά. Ψεκάστε, σκουπίστε. Και πάμε να φάμε. Θα φύγουμε στις 29 Μαρτίου του επόμενου έτος, αλλά οποιαδήποτε ψευδέστηση ε, έχουμε ότι θα είμαστε ανεξάρτητοι, νομίζω ότι ε, διασπάστηκε. Ο πρόεδρος Μακρόν ε, σηκώθηκε και αποφάσισε να μας απειλήσει. Καταλαβαίνω ότι οι Γάλλοι παίρνουν 90% των αλευμάτων στις θάλασσές μας και εμείς έχουμε μόνο 10%. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε στο έλεό σα τα επόμενα χρόνια και πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική διακήρυξη δεν μας δώσετε τίποτα σε αυτήν. Δεν χρειάζεται να μας δώσετε τίποτα και γι' αυτό λοιπόν θα αποτύχει και δεν θα περάσει από, από τη Βουλή μας και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Κύριε Μπαρνιέ, λέτε ότι είναι η μοναδική δυνατή λύση, η μοναδική δυνατή συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Ίσως λοιπόν να μεγαλώσουμε λίγο και να ηλικιωθούμε όλοι μας και να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο στις 29 Μαρτίου με ε, χωρίς συμφωνία στα πλαίσια του ΠΟΕ. Χρειάζεται μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει με υπεύθυνο τρόπο τα σύνορα. Είσαστε διτεθειμένος για κάτι τέτοιο, κύριε Μπαρνιέ, γιατί φαίνεται ότι θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται να το επικυρώσει όλα αυτά το Βρετανικό Κοινοβούλιο και δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο Βρετανικό λαό πριν από δύο χρόνια αποφάσισε να καταλήψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σεβαστούμε την κυρίαρχη του ετοιμιγορία. Ε, για την ομάδα μου, την, την Ευρώπη τη Ελευθερία των Αθνών, ο σεβασμό τη ελευθερία κάθε έθνου είναι θεμελιώδη αρχή. Οπότε οποιαδήποτε αμφισβήτηση του Brexit ε, που κατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα εκδώσει απόφαση 4 Δεκεμβρίου. Κανένα όμως δικαστήριο κατά τη γνώμη μου δεν, δεν έχει τη δικαιοδοσία για να αμφισβητήσει τα αποτέλεσματα ενός δημοψηφίσματος. Αυτό το κατάλαβε το Γαλλικό Συνταγματικό Δικαστήριο και δεν ελέγχει δημοψηφίσματα. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να θετήσει την ίδια θέση. Γιατί αν ερμηνεύσει το άρθρο 50 της Συμφωνίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσμενώς για τον Brexit, θα πρέπει να αντισταθούμε σε τέτοια απόφαση δικαστική. Γιατί η κυριαρχία δεν είναι ε, κάτι που υπάγεται στη συνθήκη ή στην υποκειμενικότητα των δικαστών. Είναι μια μετανομική ε, κατάσταση που επιτρέπει σε κάθε χώρα να διαλέξει ελεύθερο το πεπρωμένο του. Ζήτω ο Βρετανικός λαός, ζήτω και τον Brexit. Ο κύριος Κάρβερ. Ε, η Άγγελα Μέρκελ είπε το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το πιο σημαντικό για μας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να μην μπορεί να αποφασίζει μονομερό πότε θα σταματήσει η Τελωνιακή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να βρούμε από κοινού αυτό το χρονοδιάγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξακολουθούν να μας ε, ε, ανέλαβαν τον έλεγχο από το 1973 και συνεχίζουν ε, με το 2018 με τη συμφωνία προδοσίας που είναι το Brexit, η συμφωνία για το Brexit. Χάσαμε την ελευθερία μας και παρόλα αυτά, παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του 2016 ε, μας υπενθύμησαν ότι ο Βρετανικός λαός τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος θέλουμε να ανακτήσουμε στη Βρετανία την εθνική μας κυριαρχία. Οπότε όταν, είπαμε, όταν ακούσαμε ότι η κυριαρχία δεν είναι κάτι που τη, που δίνουν αλλά πρέπει να την παίρνουμε. Και σίγουρα οι Βρετανοί πολιτικοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η ιστορία θα τους κρίνει. Και πιστέψτε μου, θα τους κρίνει πολύ αρνητικά. Κυρία Πρόεδρε, πολλοί ε, ε, φιλοευρωπαίοι συνάδελφοι μου παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο κακή είναι αυτή η συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το Βασίλειο. Και σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε τόσο μονομερή βάση. Ευχαριστώ. Και τώρα... Ε, για να ολοκληρώσουμε, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Brexit, ο Μισελ Μπαρνιέ. Κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση κυρίως τον ε, Κίφερ Χόφστα, τον Έλμαρ Μπρόκ, τον κύριο Γαλτιέρη, τον κύριο Λάμπερ, την κυρία Τσίμερ που εκ μέρου ε, των πολιτικών τους ομάδων εξέφρασαν την ε, αναγνώρισή τους και την εκτίμησή τους για το έργο μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρόκειται όμως για ένα συλλογικό έργο. Δεν ήταν μοναχικό ή προσωπικό ατομικό έργο. Ήταν ένα συλλογικό έργο. Και με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, γιατί γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα διατέλεσα κάποια στιγμή και ευρωβουλευτή. Φυσικά ε, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, φάνηκε πόσο σημαντικό ήταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί ως ε, ειδικευμένο εμπειρογνώμονας υπέρ αυτής της Ένωση ενότητας μεταξύ των 27 χωρών μελών και μεταξύ των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων. Και σίγουρα θα, θα μεταφέρω τις ευχαριστίες σας ε, στην ε, Σαμπίν Βεγιάντ, στο Σεφάν και σε, όλο το επιτελείο μου που νομίζω ότι δικαίως ε, έλαβε αυτά τα εύσχημα και θα τα εκλάβει ως ενθάρρυνση. Είναι πραγματικά, ήταν πολύ σοβαρή στιγμή και πολύ θλιβερή στιγμή όπως είπατε όλοι η συμφωνία. Κύριε Φαράζ, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι φιλονικίες. Ποτέ δεν είχα εμπλέκει σε τέτοια ε, διαμάχη και θα το κάνω σήμερα. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, υπέρ της συζήτησης με όλους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όπως είπε η Γκαβρίλα Τσίμερα, μένει και η στιγμή της κύρωσης. Και τους επόμενους μήνες θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, γιατί τις χρειαζόμαστε με άλλες νομικές βάσεις βέβαια για την εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα πρέπει να επαγρυπνούμε, όπω μα υπενθύμησε και ο Γκίφερ Χόφστατ, ε, να επαγρυπνούμε για την εφαρμογή των διατάξεων τη συνθήκη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτέ οι εγγύσει που δόθηκαν, αυτά τα εχέγγυα, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και να διασφαλιστούν, ώστε οι πίκοοι και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου να μην πληγούν και να είναι εφαρμογή των δικαιωμάτων όσο πιο απλή γίνεται. Λοιπόν, επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα. Αυτό ακούσαμε και είναι απαραίτητο γιατί η συμφωνία δεσμεύει το μέλλον της Ένωσης και δεσμεύει το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και φυσικά ε, εκφράζω το μεγάλο σεβασμό μου προς τη δημοκρατική συζήτηση που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, λόγω του πολιτισμού της, του, πολιτισμού του, της ιστορίας του, την, της ιδιαιτερότητας των τραγικών στιγμών που περάσαμε ε, τον 20ο αιώνα, ε, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ελληνική μου. Και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ ποιοτική διπλωματία και είναι μια χώρα που αναφυσβήτητα χρήζει μεγάλου σεβασμού. Και ε, πραγματικά θέλουμε μια αγνής εταιρική σχέση που είναι εταιρική σχέση άνευ προηγουμένου, δεδομένου του εύρου της συνεργασίας και γι' αυτό θα εμπεδώσουμε τη συμμαχία μας ε, και όπως κάνουμε και με τις άλλες χώρες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ή διμερός για να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση και σε ένα άλλο πλαίσιο και να σφυριλατήσουμε και να εμπεδώσουμε και τη φιλία μας με, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Φαράζ, στις διαπραγματεύσεις μερικές φορές με ρώτησαν αν θα κάνουμε υποχωρήσεις, παραχωρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε στο πνεύμα ε, ο νικητής, ποιος είναι ο νικητής, ποιος είναι ο χαμένος. Το Brexit ε, μόνο χαμένους έχει. Το Brexit δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία. Θα λάβουμε υπόψη φυσικά την κυρίαρχη, την κυρίαρχη απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριε Λεμπρετών. Σεβόμαστε αυτή την κυρίαρχη απόφαση της πλειοψηφίας των Βρετανών πολιτών και θα την εφαρμόσουμε με βάση τις ενδείξεις, τα αιτήματα και τις κόκκινες γραμμές που έθεσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τον 1,5 χρόνο που εργαστήκαμε, τις διαπραγματεύσεις είχαμε με την κυβέρνηση της Τερέζας Μέη. Και ε, φυσικά, ανάλογα με αυτά που λέγαμε, έγιναν κάποια σημεία δεκτά και κάποια όχι. Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το δημοψήφισμα, να αποχωρήσει από την ενιαία αγορά. Γιατί δεν θέλετε πια να σεβαστείτε το, το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν θέλετε να σεβαστείτε την ελεύθερη, την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων. Δεν θέλετε να δεχτείτε το ρόλο του ΔΕΚ. Δεν θέλετε να πληρώσετε και θέλετε μια κοινή, ε, δεν θέλετε μια κοινή εμπορική πολιτική και αυτό δεν θέλετε και την Τελωνιακή Ένωση. Αυτή είναι, αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές σας και τις σεβόμαστε. Αλλά και εσείς θα πρέπει να σεβαστείτε τη δική μας αποφασιστικότητα να διαφυλάξουμε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την ενιαία αγορά ήμουν και αρμόδιος επίτροπος για πέντε χρόνια και σίγουρα το Ηνωμένο Βασίλειο είχε μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της ε, ενιαίας αγοράς και παρόλα αυτά την εγκαταλείπετε γιατί δεν θέλετε πια να σεβαστείτε τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και θα έλεγα και προς τον Τζέφρι Βαν Garden, ότι δεν είναι ακαμψία αυτή, δεν είναι εναλλεστικότητα και το λέω με κάθε σεβασμό. Είναι υπευθυνότητα. Έχουμε το καθήκον και την υπευθυνότητα και την ευθύνη να εργαστούμε υπέρ μιας έφτακτης αποχώρησης, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ το Brexit δημιουργεί μια ανασφάλεια. Μόνο μια ομαλή και έφτακτη αποχώρηση θα δημιουργήσει τις βάσεις και τα θεμέλια για την εμπιστοσύνη και μια ε, ε, ευρυθή και ευρύ εταιρική σχέση στην οποία προσβλέπουμε όλοι. Αυτά ήθελα να πω. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν γιατί αποχωρείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίσατε να αποχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που μας λυπεί, που μας ε, λυπεί ιδιαίτερα, γιατί ήταν αρνητική αυτή η διαπραγμάτευση χωρίς προστιθέμενη αξία. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την αίσθηση της ε, θλίψης. Κάτι που δεν μας εμποδίζει να είμαστε διαυγείς και νυφάλοι για να αντλήσουμε και τα διδάγματα αυτού του Brexit. Όπως είπαν ε, και ο Έλμαρ και ο Γκί, θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την ετοιμιγορία αυτή του Βρετανικού λαού από το δημοψήφισμα και ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες και στα αιτήματα, στις αγωνίες μερικές φορές των Ευρωπαίων πολιτών. Και πραγματικά προσπαθήσαμε να σφυριλατήσουμε αυτή την ενότητα που ζήτησαν και οι ηγέτες των χωρών μας σε αυτή την δύσκολη, κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, γιατί από όλε τι πλευρές βαλόμαστε ανατολικά, δυτικά. Ε, θελήσαμε λοιπόν να διαμορφώσουμε αυτή την ενότητα μεταξύ των 27 χωρών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και σίγουρα ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς και ε, πολύ ανηφορικός. Ε, περιμένουμε στις 11 Δεκεμβρίου την ψηφοφορία και τη διαδικασία κύρωσης από τη Βρετανική πλευρά για αυτή τη συμφωνία που είναι η μόνη, η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Και ελπίζω ε, ότι αυτή η ενότητα που διαμορφώσαμε σε αυτή την αρνητική συγκυρία, την αρνητική διαπραγμάτευση, ε, να καταφέρουμε να τη θέσουμε στην υπηρεσία ενός θετικού προγράμματος. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ, κύριε Μπαρνιέ. Και εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Πρόεδρου Ταγιάννη για την συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο, για το πνεύμα διαφάνειας και πάνω απ' όλα την υπομονή που επιδείξατε σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όρους ε, προσωπικούς επιτρέψτε μου να αναφερθώ η λέξη rubbish βλακίες αηδίες ακούστηκε αρκετές φορές δεν νομίζω ότι ήταν σωστό ε, το ότι χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις μέσα στην Ολομέλεια Νομίζω ότι τα όσα ακούσατε αγαπητοί συναλφιακτός μικροφόνου ε, σας δίνουν να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης προβλέπει τη συζήτηση με δηλώσει του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμασία διακυβερνητική διάσκεψη του Μαράκε που θα πραγματοποιηθεί στι 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση και εκ μέρου του Συμβουλίου θα λάβει το λόγο κυρία Ετστάτλερ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αξιότιμη κυρία Υπατή εκπρόσωπε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για άλλη μια φορά το θέμα, ύστερα από τη συζήτηση που έγινε στο Στρασβούργο νωρίτερα αυτό το μήνα πιστεύω ότι και με την παρουσία της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου στο Μαρακές αποδεικνύεται πως η μεγάλη σημασία αποδίδεται σε αυτό το θέμα, δηλαδή την ε, προαγωγή μιας συμφωνίας για την οργανωμένη και νόμιμη μετανάστευση μετά το πρώτο σχέδιο της, ε, του συμφώνου αυτού ξεκίνησαν οι συζητήσεις ε, και στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής αλλά και υπό την ε, Αυστριακή Προεδρία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξεκίνησαν ταυτόχρονα και οι συνομιλίες στην Νέα Υόρκη μετά την υιοθέτηση της διακήρυξης για τους μετανάστες και πρόσφυγες η Ευρωπαϊ... του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει ενεργά στην διατύπωση ενός προσχεδίου, ενός πρώτου σκαρυφήματος αυτού συμφώνου. Το Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, δεν έχει καταλήξει κοινή θέση για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ή τείνουν να αποφασίσουν ε, να προχωρήσουν προς μια κοινή θέση. Η διακυβερνητική διάσκεψη του Μαρακές μετά την υιοθέτηση από τα Ηνωμένα Έθνη και την ε, Γενική του Συνέλευση αυτού του συμφώνου ε, κηρύττει την έναρξη της ε, φάσης εφαρμογής. Έτσι λοιπόν, συνεργασία με τρίτα κράτη παραμένει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Ο διάλογος υποστήριξη προσφέρουμε στους εταίρους μας μέσω πληθώρας μέσων συμπεριλαμβανομένου και το καταπιστεύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική αποτελούν απόδειξη αυτή της ε, προσήλωσής μας στην ε, αναγνώριση των ε, αναγκών των χωρών προελεύσεως, δια, διελεύσεως και προορισμού. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Τσιτάτλερ η Αντιπρόεδρος και η Πατή Εκπρόσωπος, κυρία Μογκερίνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τη διαρκή προσοχή που προσφέρετε στο θέμα αυτό και το έργο των Ηνωμένων Εθνών αλλά και γενικά στο θέμα της μετανάστευσης. θέμα μεγάλης σημασίας και κέριο για τη δουλειά μας και τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο σφάλματα πιστεύω πρέπει να αποφύγουμε όταν συζητούμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Και άλλο ένα που θα αναφέρω μετά. Το πρώτο σφάλμα θα ήταν να θεωρήσουμε ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ εθνικών συμφερόντων και της ιδέας ενός παγκόσμιου συμφώνου. Το αντίθετο ισχύει όμως. Εάν είναι εθνικό μας συμφέρον η διευθέτηση, η ρύθμιση της ε, μετανάστευσης, κάτι το οποίο φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε, πως ισχύει δηλαδή να καταστεί πιο ανθρώπινη, νόμιμη, ε, τότε οπωσδήποτε χρειάζεται ένα παγκόσμιο σύμφωνο. Δεύτερο λάθος θα ήταν να θεωρήσουμε ότι η μετανάστευση είναι αντιπαράθεση μεταξύ βορρά και νότου της υφηλίου ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. Αλλά και πάλι το αντίθετο ισχύει. Σα αναφέρω και μόνο το εξή ότι πολλές χώρες, οι περισσότερες χώρες είναι ταυτόχρονα χώρες προελεύσεως, διέλευσεως και προορισμού, όπως οι παραδείγματι χώρες της Αφρικής. Και όπως είπα, δεν ισχύει η αντιπαράθεση μεταξύ βορρά-νότου ή νότου-βορρά, γιατί όλοι έχουμε κοινό συμφέρον να διαχειριστούμε σωστά τη μετανάστευση, συμφέρον για την επένδυση, για τις βιώσιμες επενδύσεις στις χώρες προελεύσεως και την εξασφάλιση νόμιμων οδών διελεύσεων και κινητικότητα. Όσο πιο νωρί λοιπόν αντιληφθούμε ότι η εταιρική σχέση και η συνεργασία είναι αυτό που πράγματι χρειαζόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί σε αυτό όλοι βρισκόμαστε μέσα στην ίδια κατάσταση. Καμία χώρα μόνη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Ε, και όλες οι χώρες έχουν ε, συμφέρον να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο κατά τρόπο τακτό. Και επίσης υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εθνών Πανκιμούν για την επαναφορά στην ημερήσια διάταξη του θέματος όπως άλλωστε είχε ξεκινήσει το 2016 τη Γενική Συνόλευση και την υιοθέτηση της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα για τους πρόσφυγες και για τη μετανάστευση σημαντικά επιτεύγματα για μας τους Ευρωπαίους διότι στο επίκεντρο μιας μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη και τονίζω στην Ευρώπη γιατί πρέπει να τονίσω ότι οι μεταναστευτικές κρίσεις ανα πάσα στιγμή υπάρχουν και σε οδήποτε σημείο του κόσμου καταγράφονται αλλά μετά από αυτή την σύνοδο του 2016 και στο επίκεντρο όπως είπα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης η Ευρώπη, εμείς καλέσαμε την Ευρωπαϊκή, τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει εταιρικέ σχέσεις και να χορηγήσει μια θετική ανταπόκριση και εδώ ακριβώς ήταν και η ρίζα από την οποία ξεκίνησε το Παγκόσμιο σύμφωνο ε, από ε, πρώιμη φάση έλαβε μέρο η Ευρωπαϊκή Ένωση στι συνομιλίε και διαπραγματεύσει για το Παγκόσμιο Σύμφωνο εξ αρχή ε, με τρόπο ενεργό για να καταλήξουμε σε, στι σαφέ αυτέ κοινέ θέσει που έχουμε μπροστά μα και έτσι μπορέσαμε να προωθήσουμε ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο που σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει του ευρωπαϊκού στόχου, κάνοντα σεβαστέ όλε τι ανησυχίε μα και όλα τα μελήματά μα. Και ξέρω ότι ο Επίτροπο Τηλιανίδη στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδε περίπου είπε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξέφρασε τη λύπη τη Επιτροπή για το γεγονό ότι υπάρχουν χώρε στο Συμβούλιο που δεν δέχονται και δεν υποστηρίζουν το Παγκόσμιο Συμφώνιο για τη Μετανάστευση. Πιστεύουν ότι τα συμφέροντα όλων των κρατών εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο εφόσον προωθηθεί αυτό το σύμφωνο, γιατί αποτελεί μια βάση για διεθνή συνεργασία και διάλογο, βάση η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Βάση την οποία εμεί ζητήσαμε. Διάλογο και συνεργασία που ήδη εγγράφονται στην, ε, στο πλαίσιο των και τη βάση των αποτελεσμάτων που χρειάζεται ακόμη βέβαια να, ε, να εδρεωθούν και που εμείς προκαλέσαμε μετά όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή εναλλακτικέ οδοί, εναλλακτικέ για τους ε, πρόσφυγες, αντιμετώπιση ποινική των διακινητών, ε, επαναπροωθήσεις, μέτρα δηλαδή για ομαλή επαναπροώθηση, όλα αυτά που θα ήταν μέτρα που θα οδηγούσαν σε εταιρικέ σχέσει, συνεργασία, σε, σε πνεύμα αμοιβέ κατανόηση και εμπιστοσύνη μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά είναι κομμάτι του παγκόσμιου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε παρεξηγήσει και θέλω να υπογραμμίσω μία. Είναι αυτονόητο για μένα, αλλά ίσω θα πρέπει, δεδομένου ότι έχουν προχωρήσει, όπω έχουν προχωρήσει συζητήσει σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να το τονίσω. Νομικά δεσμευτικό δεν είναι το σύμφωνο αυτό και νομίζω ότι πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε εξ αρχή και να τονίσουμε ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό το σύμφωνο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, να γεννήσει αδίποτε ένομη συνέπεια για τα συμβαλόμενα μέρη. Είναι απλώς ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών, προτάσεων, συστάσεων για το τι μπορούν να κάνουν σε τρόπο, με, με τρόπο συνεργατικό, σε διεθνές επίπεδο. Τα κράτη-μέλη αποτελεί ένα πλαίσιο, προσφέρει ένα πλαίσιο και έτσι αποτελεί και, στη, και χτίζει πάνω σε αυτή βάση τη βάση δηλαδή τη εθνική κυριαρχία και τη ε, κυριαρχία των κρατών να προσδιορίσουν μόνα του την μεταναστευτική του πολιτική. Παράλληλα όμω αποτελεί ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα πλαίσιο το οποίο εμεί οι Ευρωπαίοι ζητήσαμε. Θα συνεχίσουμε βέβαια να προσπαθούμε ε, και να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη διαχείριση μετανάστευση όπω γίνεται αυτή τη στιγμή ήδη από πλευρά Ευρωπαϊκή με βάση και τι παγκόσμιε τάσει, ε, όπω αυτέ περιγράφονται από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Δεν θα διακόψουμε τη συνεργασία μα με τη Διεθνή Οργάνωση μετανάστευση. Θα συνεχίσουμε θα προχωρήσουμε και μετά το σύμφωνο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν ε, και όλες οι χώρες να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις αποτελεσματικές. Θα ξεκολουθήσουμε να υποστηρίσουμε εταιρικέ σχέσεις και διμερείς και πολυμερείς στον τομέα της ε, μετανάστευσης χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη ε, σημαντική αυτή τη σημαντική βάση συνεργασίας που είναι το Σύμφωνο Μετανάστευσης και που ε, εκφράζει, όπως είπα, την ευρωπαϊκή προσέγγιση μετανάστευση. Κοινή δουλειά δική μας, συμβολή δική σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι απαραίτητη, απαραίτητα στοιχεία για τη Σύνοδο του Μαρακέσου. Ε, θα ηγηθεί τη Ευρω... Ευρωπαϊκή ε... Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Χαίρομαι που βλέπω ότι θα υπάρχουν και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου στη κυβερνητική αυτή διάσκεψη. Χαίρομαι και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει κέριο ρόλο να διαδραματίσει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον, για την προσήλωση, για την στατευμένη εργασία στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για να μην λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ζόφκο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, ως μέλος της Επιτροπής ΦΕΤ και ΔΕΒΕ, φυσικά γνωρίζουμε πόσες αιστείες έναπλων υπάρχουν και ε, που έχουν οδηγήσει στην έξοδο πολλών ε, πολιτών από τις αιστείες τους. Το 2015 είδαμε πως αρκεί μία μόνο σπίθα για ε, να απειλήσει την ειρήνη στα Βαλκάνια και να ξεκινήσει ένα μεταναστευτικό ή προσφυγικό κύμα. Η Κροατία που έχει τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα με τα Δυτικά Βαλκάνια το γνωρίζει καλά. Η Ιταλία και η Ισπανία με τα θαλάσσια σύνορα προς την Αφρική ήταν περισσότερο εκτεθειμένες στο προσφυγικό κύμα και δεν μπορέσαμε να ορθώσουμε ε, τύχη. Και σίγουρα ε, δεν θα πρέπει ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα αυτό το πρόβλημα, αλλά να επιδιώξουμε παγκόσμιες λύσεις και συνεργασία. Λυπάμαι που το σύμφωνο, ε, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ε, δημιουργεί διχασμούς ε, και προβλήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να εγκρίνουμε αυτό το σύμφωνο και μάλιστα ήμουν από τους επικεφαλείς των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του ΕΛΚ. Ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή για να υποδεχθούμε τους πρόσφυγες με ανθρώπινο τρόπο. Ευχαριστούμε την κυρία Ζόφκο. Ένα λεπτό έχει η κυρία Αξιότιμοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση ζητήθηκε γιατί πολλές ε, ευρωπαϊκές ε, κυβερνήσεις αποφάσισαν να αποχωρήσουν από αυτή τη συμφωνία και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και να Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτή τη συμφωνία με μεγάλη πλειοψηφία, γιατί πρόκειται για μια συμφωνία η οποία τονίζει και βάζει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι η διεθνή συμφωνία υπονομεύει την επικυριαρχία των κρατών και ότι προμηνεί την κατάπτωση της δυτικής του δυτικού πολιτισμού, γιατί τέτοια ακούμε και συχνά στι συζήτησει στη Σλοβανία. θεωρώ ότι πρόκειται για πραγματικά σχόλια, πρόκειται για πολιτικές δηλώσει. Βασίζεται η συμφωνία αυτή στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ένωμη Τάξη, στον καταμερισμό των ευθυνών και των υπευθυνότητων. Εγώ επέστρεψα από τον Ήγηρα, όπου ο κόσμος καθημερινά αγωνίζεται, πολεμάει για μια αξιπρεπή ύπαρξη για τους ε, φυσικούς πόρους που εκμεταλλεύεται ο δυτικός κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαγιόν και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Βίστησεν. Συμφωνία του Μαρακέσα αποτελεί ένα συνοθήλευμα φιλελεύθερων ιδεών που έχει φέρει την Ευρώπη στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα γιατί δεν κατανοούμε το φαινόμενο της ε, μη ρυθμισμένης μετανάστευσης. Ποια είναι η λύση λοιπόν ε, για το θέμα αυτό αν ε, πιστέψουμε τον ΟΗΕ να δώσουμε πιο πολλά δικαιώματα, να προωθήσουμε ακόμη πιο πολύ μετανάστευση και όχι την επιστροφή των μεταναστών. Είμαστε από τα κράτη-μέλη που δεν θέλουμε να υπογράψουμε μια τέτοια τρελή συμφωνία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι και πολλές άλλες τέτοιες χώρες, ε, η ΙΠΑ, η Αυστραλία. Ωστόσο, έχουμε πάρει την απόφαση καλούμε την κυβέρνησή μας να μην ακολουθήσει την τάση για να υποστηριχθεί και να υπογραφεί αυτή η τρέλα από το Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαρτζεντίνη τώρα για ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, πρόεδρε η σχιζοφρένεια επικρατεί. Εδώ ακούμε την Αυστριακή κυβέρνηση που μιλάει εξ ονόματος του, της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και μιλάει με ωραία λόγια, αλλά δεν θέλει να τα υποστηρίξει αυτά η Αυστριακή κυβέρνηση. Και από την άλλη μας μιλάει η κυρία Μοργκερίνη, η οποία εκπροσωπεί και την Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο για την Ασφαλή Μετανάστευση. Το γεγονός ότι δεν θα ακολουθούσε ο Τραμπ λοιπόν δεν ήταν ένα πάντεχο. αλλά εμείς η Ευρώπη της ήπιας δύναμης, εμείς υποτίθεται ότι θα δείχναμε σε όλο τον κόσμο ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με μια συμφωνία για να φροντίσουμε τα παιδάκια των μεταναστών να, να πάνε στο σχολείο. Τα παιδιά να μην βρίσκονται χωρίς έγγραφα, να μπορούν να έχουν μία ύπαρξη. Ήταν η δική μας στιγμή να φροντίσουμε να μην μας κρατούν όμοιρο οι κρίσεις, ε, οι μεταναστευτικές του 2015. Και τι κάνουμε αντί αυτού, παίζουμε ιστορικά παιχνίδια και ξεχνάμε ότι θέτουμε πρότυπα τα οποία ισχύουν και για την Αφρική αλλά και για την Ασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρτζεντίνη. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά ανήκουστο κάποιες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω ξενοφοβία ή ρατσισμού να αποσύρονται από το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Και στην ε, αριστερά έχουμε προβλήματα με το Σύμφωνο του Μαρακέ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιοι στόχοι ε, και διαδικασίες για να διαχειριστούμε τη μετανάστευση. Δεν είναι πρόβλημα η μετανάστευση. Η εκμετάλλευση των μεταναστών είναι πρόβλημα και αυτό το βλέπουμε ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θέλουμε μια εξωτερική πολιτική και να αποτρέψουμε και το εμπόριο όπλων ή το λαθρεβόριο ανθρώπινων όντων. Θα πρέπει να έχουμε πραγματικά κοινέ δράσεις για να οδηγηθούμε σε αυτά αποτελέσματα. Αλλά να δούμε ε, ότι και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μπει σε στραβό δρόμο, γιατί πρώτα δεν διορθώνουμε τα του οίκου μας. Ε, ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να υποδεχθούμε με αξιοπρέπεια τους μετανάστες. Ε, έχουμε πολλά σημεία που θα πρέπει να διορθώσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση. Επίσης, ε, είναι πραγματικά επονίδιστο το ότι πολλοί δαιμονοποιούν τους μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόιτεν, ένα λεπτό. Πρόεδρε, για άλλη μια φορά μιλούμε για Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, γιατί η πράσινο-αριστερή ουτοπική πολιτική ελπίζει να απο να προκύψει από το Κοινοβούλιο ένα θετικό μήνυμα για την διευκόλυνση τη μετανάστευση. Το αντίθετο όμω θα συμβεί. Η Ιταλική κυβέρνηση χθε αποφάσισε να μην υποστηρίξει το σύμφωνο μετανάστευση. Έτσι, όλο και πιο μακροσκελή στο κατάλογο των κρατών αικαιών που στρέφονται κατά αυτή του παράλογου θεματολογίου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Αυστραλία, το Ισραήλ, η από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσοχία, η Σλοβακία και βλέπουμε ότι κρίνεται μια κρίση και στη Γερμανία ακόμη που θα δώσει απαντήσει σε αυτόν τον παραλογισμό της κυρία Μέρκελ που θέλει την ε, χώρα μα να καταστεί κέντρο μεταναστευση. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε αυτό το σύμφωνο. δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα. Αυτά τα fake news πρέπει να τα σταματήσουμε και πρέπει να σταματήσουμε την πορεία αυτού του συμφώνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μότιν. Βιλίμσκι, πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ξεκινά μια όμορφη μέρα, μια καλή μέρα σε ένα μακρινό κράτος όπου δεν πρόκειται, ε, με ένα ακόμα κράτος το οποίο δεν πρόκειται να υποστηρίξει το σύμφωνο. Ο Σαλβίνη αποφάσει εκ μέρου Ιταλία ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσει στο σύμφωνο όπω και πολλέ άλλε χώρε. Ηνωμένε Πολιτείε, Αυστραλία, ε, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία ε, όλο και περισσότερε είναι οι χώρε και αν δείτε ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι των ΗΕ, καμία σχέση δεν έχουν με το σύμφωνο μετανάστευση. Οι κύριοι στόχοι είναι ο αφοπλισμό, η ειρήνη, η ασφάλεια για του πολίτε. Αυτή είναι η στόχη των ΗΕ. Αλλά έχουν μετατραπεί Ηνωμένες, ε, τα Ηνωμένα Έθνη σε κάτι άλλο και δεν έχουν οπωσδήποτε καθόλου στόχο ιδρυτικό την διευθέτηση τη μετανάστευση ή την παρισύφρηση σε αρμοδιότητες και εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν ότι πια ξυπνούν και το βλέπουν όλο και προς τώρα κράτη και γι' αυτό κανένας πλέον δεν θέλει να προσχωρήσει αυτό το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Βιλίμσκι. Κύριε Φόικτ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με ξαφνιάζει κυρία Μογκερίνη που λέτε ή τολμάτε να λέτε ότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη το σύμφωνο τα κράτη ύστερα από τέσσερα χρόνια καλούνται να επαληθεύσουν εάν τα μέτρα του συμφώνου έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Και Μπορεί βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι η νέα λέξη της μόδας και η μαγική λέξη θα είναι η ενσωμάτωση, η συμπερίληψη στις κοινωνίες, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να προκύψει από τη Σύμβαση των Εθνών για τους πρόσφυγες, δηλαδή ότι μπορεί αυτοί οι μετανάστες ε, που μπορεί να ε, μην κινδυνεύουν από πόλεμο στις χώρες τους θα πρέπει να επαναπατρίζονται, σταματάει ως επιλογή και πλέον η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση γίνεται η μαγική λέξη και άρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, έχουν βρει την λύση πολλοί λαοί και δεν πρόκειται να υπογράψουν το σύμφωνο μετανάστευσης. Πιστεύω ότι και οι μετανάστες οι ίδιοι δεν έχουν ε, ε, δει θετικό τίποτα για το μέλλον τους από αυτό το διάκοψε ο Πρόεδρος. Κύριε Φόικτ, ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κοράτσα μπίλτ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Μογερίνη, το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι σημαντικό γιατί αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση είναι μια παγκόσμια ε, πρόκληση και χρήζει παγκόσμια ε, λύση και αλληλεγγύης. Και οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν περισσότερες μετακαταστάσει. Λυπάμαι που ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Παγκόσμιο Σύμφωνο, αλλά το χειρότερο είναι ότι και χώρε μέλη αποχώρησαν. Γιατί το να λέμε γυρίστε σπίτι σα και παραμείνετε εκεί δεν είναι λύση. Κανένα κράτο δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και παγκόσμια συνεργασία. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση. Γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε στην Ευρώπη με τρίτε χώρε για την πρόληψη, για την καταπολέμηση τη ε, εμπορία ανθρώπων και ε, και την επιστροφή. Και επίσης θα πρέπει μακροπρόθεσμα να επενδύσουμε στην Αφρική. Ήμουν στη, στον Ήγηρα και στο Αγκαντές μαζί με την αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χάρη στην αποτελεσματική δράση μειώσαμε τη μετανάστευση, σώσαμε ζωές, καταπολέσαμε τη λαθροδιακίνηση, χάρη σε περισσότερη και ισχυρότερη εταιρική σχέση με την Αφρική. Και δυστυχώς διακόπτει το μικρόφωνο της κυρίας Κόρα Ευχαριστώ κύριε Κόρατσα Μπίλτ. Μιούλερ, ένα λεπτό. Ένα τέτοιο παγκόσμιο σύμφωνο αποτελεί μια σημαντική συμβολή σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες απαντήσεις που χρειαζόμαστε για την μετανάστευση. Αποτελεί ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δημιουργεί σαφείς κανόνες και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα σε χορήγηση ασύλου δεν το αμφισβητεί τουλάχιστον. Είναι κρίμα λοιπόν που κάποια ευρωπαϊκά κράτη δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν όσοι απορρίπτουν τη διακήρυξη αυτή δεν ενδιαφέρονται να βρεθεί μια λύση. Ουσιαστικά θέλουν να παραμείνει πρόβλημα το ζήτημα της μετανάστευσης, γιατί από αυτό μπορούν να υποφεληθούν σε πολιτικούς όρους. Αυτό πραγματικά είναι απάνθρωπο. Και τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις θα μας πλέξουν όλους. Θα πρέπει να ταχθούμε κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ευχαριστώ κύριε Μέλλερ και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Φίτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόεδρος Μογκερίνη είπε μόλις τώρα ότι ε, το Παγκόσμιο Σύμφωνο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη. Διαρωτώ με λοιπόν 10-11 Δεκεμβρίου στο Μαρακές θα γίνει μια μεγάλη συνέλευση που θα συζητηθεί αυτό γιατί η πραγματικότητα είναι ότι για τη μετανάστευση που είναι μεγάλη αποτυχία των κρατών τα τελευταία χρόνια παίχτηκε ένα σε πολιτιστικό σε επίπεδο νοοτροπίας δηλαδή αλλά και σε πολιτικό επίπεδο παιχνίδι και είναι καλό να μην συμμετέχουμε σε μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία έχει τελείως αβέβαιη έκβαση και προ τελευταία ανάλυση το μόνο που κάνει είναι να ε, προβάλλει μια πολιτική δράση στοχευμένη, η οποία όμως σημαίνει απλώ ότι συνεχίζουμε σε ένα λάθο δρόμο. Μιλήσανε πολλοί συνάδελφοι για την αποχώρηση τη Ιταλία. Η Ιταλία χρόνια, ε, μέρες τώρα μιλάει, χάρη ακριβώ και στην παρέμβαση τη Τζόρτζια Μελώνη, των Φρατέλε Ιταλία, αδελφών τη Ιταλίας, που συμμετέχει και στηρίζει μια κυβέρνηση ο Σαλβίνη είπε ότι δεν πρόκειται να πάει, ενώ ο Κόντε, ο Πρωθυπουργό, είπε ότι θα πάει στο Μαρακέ. Ε, αυτή ήταν η αβεβαιότητα που είχε η Ιταλία. Αλλά εμεί από του Φρατέλη τη Ιταλία αγωνιζόμαστε ώστε να, ώστε να μην συμμετάσχει η Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ, Μπορκέτσιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ δεν θα παραθέσω τα λόγια του Σαλβίνη, αλλά του Πάπα Φραγκίσκου που, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είπε ότι η Ευρώπη, αν μπορέσει να δώσει αντίσει συγκεκριμένε για την πολιτιστική τη ταυτότητα και την την προάσπιση του δικαιώματος για υποδοχή αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών που βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς στις ίδιες τους τις χώρες όμως. Πέραν των όσων φαίνεται να διεκδικεί ο πρόεδρο Σταγιάννη με τη μορφή κάποιου νέου σχεδίου Μάρσαλ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα λόγια του Πάπα. Ε, μετά μας λέτε ότι πρέπει να έχουμε την εθνική κυριαρχία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να υποτασσόμεθα στις διεθνείς συνθήκες, άρα είναι κάπως περιορισμένη η εθνική κυριαρχία. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπνεόμεθα από εκείνους που έχουν μια κάποια ιδέα για την Ευρώπη, όπως ο Άγιος Πατήρ. Αν δεν το είχε πει ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος, εγώ θα είχα σταματήσει δεν θα συνέχιζε αυτό το επιχείρημα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και το επιχείρημα της τελική κυβέρνησης, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ευαίσθητοι ως προς τα δικαιώματα εκείνων που προσπαθούν να διαφύγουν από διώξεις κτλ. Αλλά και εκείνους, εκείνων που θέλουν να καταδικάσουν την ε, προδιακόπτη ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο και τώρα η κυρία Κέγκε για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα μεταβώ στο Μαρακές με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο προσφέρει μια παγκόσμια απάντηση στο θέμα της μετανάστευσης αποτελώντας συνέχεια της δικής μας της δουλειάς για την επίλυση με τρόπο πλήρη ολικό ε, ολοκληρωμένο καλύτερα του προβλήματος μετανάστευση Είναι πολλές οι χώρε δυστυχώ οι οποίες έχουν αποφασίσει να υπονομεύσουν την διακυβερνητική διάσκεψη και πάνω από όλε η δικιά μου χώρα, η Ιταλία που λέει και θέλω να του πω πηγαίνετε, πηγαίνετε στο Μαρακές, ελάτε, ελάτε μαζί μου, ελάτε με εμά, γιατί το Μαρακέ σημαίνει όχι μόνο λύσει για μια πιο ασφαλή ε, και σταθερή μετανάστευση αλλά και αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες. Μην μείνετε στο περιθώριο της ιστορίας. Η ιστορία αυτή είναι, η ιστορία τώρα γράφεται, δεν θα σταματήσουν μεταναστευτικές ροές, θα συνεχίσουν και πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα και να δώσουμε απαντήσεις στις βαθύτερες αιτίες μετανάστευσης και πια άλλη μια φορά θέλω να καταδικάσω την ε, υποκρισία της θελικής κυβέρνησης που προσπαθεί ενώ υποτίθεται πώ ζητά την αλληλεγγύη των άλλων για το θέμα της μετα... ο Πρόεδρο διακόπτη. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στη δικασία και βλέπουμε ότι έχουμε τις διπλάσιε αιτήσει για το λόγο σε σχέση με τον χρόνο που έχουμε. Έχουμε και ψηφοφορίε και σα ζητώ συγγνώμη αν δεν καταφέρω να ακούσουμε όλου του συναδέλφου. Ο κύριο Σφαίρη είναι πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά της παγκόσμιας αυτής της συμφωνίας των Μαρακές. Αυτή η συμφωνία δεν ε, η Αυστραλία, το Ισραήλ, και 10 κράτη-μέλη έχουν ήδη αποφασίσει να μην υποστηρίξουν τη συμφωνία αυτή. Δεν πρόκειται λοιπόν για παγκόσμια συμφωνία. 70% του σλοβενικού λαού είναι άλλωστε κατά. Και τα πολιτικά κόμματα δεν συμφωνούν από αυτό και κυρίως η ευρωπαϊκή και διεθνή κοινή γνώμη. Το κείμενο είναι κακό και δεν μπορούμε να πούμε ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Πρόκειται για ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Είμαι λοιπόν κατά της, ε, του συμφώνου αυτού, γιατί θεωρώ ότι θα είναι ακόμα χειρότερη η ρύθμιση της μετανάστευσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αντιθέσει πιο πολλούς πόρους προς την κατάλληλη Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φρόιν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτοί που απορρίπτουν το σύμφωνο μετανάστευση κατά πάσα πιθανότητα δεν το έχουν διαβάσει καν, γιατί ακολουθούν λαϊκιστικές τάσει. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το σύμφωνο για την εντολή, για παράδειγμα, για να υπάρχει μία βάση για την πολιτική μετανάστευση, απόπειρα να δίνουμε σωστές και ακριβείς πληροφορίες σε όλες τις φάσεις μετανάστευσης. Απορρίφθηκε να σώζονται ζωές και να υπάρξει συντονισμός των εθνικών και διεθνικών πράξεων διάσωσης. Απορρίπτεται καταπολέμηση των κυκλωμάτων σωστή και ασφαλή διαχείριση των συνόρων. Η κυβέρνησή μας δεν θέλει να δημιουργούνται δυνατότητες για πιο σωστή και γρήγορη και ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή των μεταναστών στα σπίτια τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φρόιντ. Η κυρία Τόμασιτς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε με ένα παγκόσμιο πλαίσιο τη μετανάστευση υπάρχει. Γιατί ότι δυστυχώς πολλές χώρες δεν σέβονται την παγκόσμια δημόσια τάξη και αυτό επηρεάζει τη μετανάστευση. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ε, α, έγγραφα, με πλαστά έγγραφα και χωρίς ε, εξακρίβωση περνάνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, πηγαίνουν σε διάφορα Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και μας απειλεί όλους. Η μετανάστευση θα πρέπει να είναι πιο ασφαλής και για τους μετανάστες αλλά και για τους συμμεταπούς. Ε, γιατί για πολλούς ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και ποιες είναι οι πραγματικές τους προθέσεις όταν έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση δεν έχουμε αυτό το πλαίσιο που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την, τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις και γι' αυτό έχουν φύγει πολλές χώρες από αυτό όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί ε, Δυστυχώ με την λύση αυτή, όπου δεν ξέρουμε ποιε χώρε θα υποδεχθούμε, αλλά ποιε αποφεύγουν το σύμφωνο, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε στον δρόμο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σόλτα. Ευχαριστώ. Αυτή η παγκόσμια συμφωνία είναι μια συμφωνία την οποία προφανώς και χρειαζόμαστε θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να επιλύσουμε πολλά προβλήματα με πιο εύκολο ε, τρόπο. Πολλά προβλήματα τα οποία μας ε, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση σήμερα. Αυτή η παγκόσμια συμφωνία θα σήμαινε μια πιο αποτελεσματική καθοδήγηση της μετανάστευσης και αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε προάσπιση των δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των κρατών μελών. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έχει πολλές και μεγάλες φιλοδοξίες αν ε, διαβάσουμε όλους τους στόχους που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια αυτή συμφωνία, θα διαπιστώσουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις, πολλές λύσεις. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να καταψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Σόλτας και στην ε, τέλος ο κύριος Επιτιδίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι ένα κείμενο όχι μόνο άχρηστο αλλά και επικίνδυνο. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζει το δικαίωμα της ε, μαζικής κινητοποίησεως και μετακινήσεως για οικονομικούς λόγους σε οποιονδήποτε από τρίτες χώρες θέλει να εισέλθει ή ακόμη και να εισβάλλει κυρίως στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του ποιος είναι νόμιμος και ποιος παράνομος μετανάστης. αυτό έχει σαν επίπτωση τα κράτη να μην μπορούν να ακολουθούν μια ανεξάρτητη εθνική μεταναστευτική πολιτική και να προστατεύουν τα σύνορά τους. επιπλέον υπάρχει κίνδυνο στο μέλλον οι μη δεσμευτικοί αυτή τη στιγμή στόχοι που αναφέρονται στο σχέδιο να γίνουν δεσμευτικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις αγκυλώσεις και την αιμονή της αριστεράς δεν θα προκαλέσει εντύπωση εάν οποιαδήποτε επίκριση για αυτό το φαινόμενο της παράνομης μεταναστεύσεως γίνει ποινικό αδίκημα. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλά κράτη δεν επιδιώχουν πλέον να γράψουν αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και τώρα να δώσουμε το λόγο λοιπόν εκ νέου στην ε, εκπρόσωπο του, ε, την κυρία Μαγκερίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι μιλώ εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή η Αυστριακή Προεδρία θα παρουσιάσει τι θέσει του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σαφή τοποθέτηση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο και όπω σα εξήγησα πρόκειται για απόρρια μια διαδικασία που ξεκινήσαμε εμεί στον ΟΗΕ. Ζητήσαμε εταιρική σχέση, συνεργασία, ένα πολιτικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο για να διαχειριστούμε μαζί τα φαινόμενα αυτά. Βάσει των όσων είχαμε ξεκινήσει ήδη με φίλου από την Ασία, την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική, από παντού. Μια βάση ναι, συγγνώμη, δεν μπορώ να σας μιλάω αν κάποιος μιλάει από δίπλα μου και δυνατά μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς τη διαδικασία αυτή στα πλαίσια του ΟΗΕ και ζητήσαμε μια πολιτική προσέγγιση, όχι πολιτικά δεσμευτική, για να δημιουργήσουμε συνεργασίες. Γιατί εμείς ως Ευρωπαίοι ανακαλύψαμε αρκετά αργά, εν παση περιπτώσει, 2015-2016, ότι χρειαζόμασταν ε, στενές σχέσεις με τις χώρες προέλευσης και προορισμού για να υποστηρίξουμε ένα κοινό σύστημα, μια κοινή προσέγγιση για την διαχείριση τη μετανάστευση, να καταπολεμήσουμε του διακινητέ, να προσφέρουμε ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε και δύσκολα θέματα, όπως είπατε κάποιοι από εσά, όπως είναι οι επιστροφές με αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό πλέον αποτυπώνεται σε ένα σύμφωνο. Ένα σύμφωνο το οποίο πέρασε από την ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Όπω σα είπα, το σύμφωνο αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τι ε, θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργασία που κάνουμε ήδη από κοινού με του εταίρου μα σε ό,τι αφορά το UIM, το UNHCR κτλ. Και να σας πω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει αντιπροσωπεία εκπροσώπουσης στο Μαρακές με τον ε, Επίτροπο Αβραμόπουλο και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον ΟΗΕ για την εφαρμογή σε τεχνικό επίπεδο, όπως ενδεχομένω να γνωρίζετε, μετά την, ε, το Μαρακές θα γίνει μια γενική συνέλευση όπου τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ θα ψηφίσουν και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ, με τις υπηρεσίες, με τους εταίρους μας σε παγκοσμίο επίπεδο για να εφαρμοστεί αυτή η ατζέντα. Γιατί είδαμε ότι στα πρώτα χρόνια της εργασίας μας, τις εργασίες μας με τις ίδιες αρχές που αποτυπώνονται στο σύμφωνο, τα αποτελέσματα ήταν φετικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, να επενδύουμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο η εφαρμογή αυτή σε ένα μη δεσμευτικό τέτοιο πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τις εργασίες με το επόμενο χρόνια. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Και ευχαριστούμε την ε, Επίτροπο κυρία Μογκερίνη. Το λόγο έχει η κυρία Έτσου Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή συζήτηση εν ώψη της ε, διάσκεψης που θα γίνει τον επόμενο μήνα και την επικείμενη έγκριση του Παγκόσμιου Σύμφωνου για τη Μετανάστευση στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή. Η μετανάστευση γενικώ, αλλά κυρίω η συνεργασία με τρίτε χώρε ε, θα εξακολουθεί να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Συμβουλίου και τη Αυστριακή Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση αυτού του στόχου και σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσετε τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες, τον προβληματισμό σας και τις σκέψεις και απόψεις σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τστέτλερ. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη έχει να κάνει με την προφορική ερώτηση με δηλώσει επιτροπή για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες. Es beginnt als Verfasserin die Frau Kollegin Κυρία έχει το λόγο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλούμε στο όνομα των άνω των 46 εκατομμυρίων γυναικών με αναπηρίες, που είναι το 16,6% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα με τη συζήτηση αυτή θα, τους, θα προβάλλουμε τις γυναίκες αυτές, θα γίνουμε ο εκπρόσωπός τους, η φωνή τους, για να μπορέσουν πραγματικά να ασκούν και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά του. Γιατί οι γυναίκε με αναπηρία είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινα πλάσματα. Είναι πολίτε που δεν θα πρέπει να τι καθορίζουμε με την αναπηρία του. Ούτε κάτι τέτοιο επιθυμούν. Και καθημερινά αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα με τι υπόλοιπε γυναίκε. Είναι σύζυγοι, μητέρε, φίλε, εργαζόμενε. Έχουν πολλαπλά ταλέντα και ικανότητε και εμπλουτίζουν την κοινωνία μα, εξασφαλίζοντα μεγαλύτερη πολυμορφία. Είναι ζωτική σημασία και η δική του συνεισφορά. Γι' αυτό και θα πρέπει να την προωθήσουμε και θα πρέπει ε, τα σχέδιά του να φροντίσουμε να γίνουν πραγματικότητα και να φογκραζόμαστε και τη δική του φωνή. Σήμερα με τη συζήτηση θα δημιουργήσουμε μια θετική και ευαισθητοποίηση για την διαφορετικότητα και θέλουμε να επιβάλλουμε την κουλτούρα της διαφοράς, γιατί αυτή η παιδεία της διαφοράς και της πολυμορφίας δημιουργεί κοινωνικά πλεονεκτήματα. Οι γυναίκε αυτέ αντιμετωπίζουν καθημερινά την πρόκληση γιατί μερικέ φορέ φαίνονται, ε, δεν φαίνονται, είναι αόρατε. Σαν να μην βλέπουν, σαν να μην ε, ε, ε ακούν. Γιατί αυτέ οι γυναίκε έχουν αναπηρίε, αλλά αποκλείονται από την ίδια την κοινωνία, γιατί μερικές φορές προσκρούν σε προκαταλήψεις που τις καθιστούν αόρατες και υποφέρουν πολλές διακρίσεις σε πολλές χώρες και σε πολλούς τομείς. Μιλούμε για παιδεία, για παιδεία χωρίς αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει ελεύθερα να συμμετέχουμε στην κοινωνία και να συμβάλλουμε στην κοινωνία αυτή με τον ίδιο τρόπο. Όταν έχουμε διακρίσεις στην παιδεία, ουσιαστικά ε, καθιστούμε ένοχο τον διαφορετικό μαθητή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε παιδεία και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς ε, για να μπορούν όλοι οι συμπολίτε μας να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς. Μόνο το 18,8% των γυναικών με αναπηρίες ε, έχουν μια θέση εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ λιγότερο ποσοστό είναι το ποσοστό των ανέργων ανδρών με αναπηρίες. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε για, για τον ψηφιακό αλφαβητισμό, γιατί οι ε, περισσότερες γυναίκες με αναπηρία είναι άνω των 60 ετών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τις ηλικιωμένε γυναίκες με αναπηρίες. Επίσης, ε, ζητούμε πλήρη και απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των ε, γυναικών με αναπηρίες σε όλους τους τομείς κοινωνίας. Δεν θα πρέπει να τις αποκλείσουμε, δεν θα πρέπει να μένουν στο περιθώριο και επίσης να κατοχυρώσουμε και να κάνουμε πραγματικό το δικαίωμα του εκλέγην και το εκλέγεσθε των γυναικών με αναπηρίες. Και έχουμε μια νομοθετική αναθεώρηση στην Ισπανία προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι στι αξίε Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θέλουμε θετικέ δημόσιε πολιτικέ για να καταρρύψουμε όλου αυτού του φραγμού στην ισότητα και κυρίω να δώσουμε απλή, αποτελεσματική και αληθινή, ακριβή πληροφόρηση στι γυναίκε για να γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Και η προσβασιμότητα είναι το προαπαιτούμενο για την ισότητα και τη συμμετοχή. Στι 8 ε, Νοεμβρίου ακούσαμε ότι Συμβούλιο και Επιτροπή συμφώνησαν γι' αυτό. Ε, τη στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία ε, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, αλλά τουλάχιστον βαίνει προς την κατεύθυνση της κατάρριψης των εμποδίων. Θέλουμε αυτή η ισότητα να γίνει πραγματικότητα. Στις, στους γυναικολογικούς ελέγχους οι γυναίκες ε, με αναπηρίες έχουν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να, να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο γυναικολογικό έλεγχο. Έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κατά της ε, ενδοικογενειακής βίας, στις υπηρεσίες ε, που παρέχουν πληροφορίες. Αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να τα καταρρύψουμε. Και ο κοινωνικός πυλώνας είναι μια ευκαιρία που μας δίνεται για να συμπεριλάβουμε και τις γυναίκες με αναπηρίες στην κοινωνία και να τους δώσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και μιλούμε και για αξιοπρέπεια. Να ξεφύγουμε από τη σιωπή, τι που υφίστανται αυτές τις γυναίκες Μία στις τρεις γυναίκες με αναπηρίες ήταν ή θα ε, είναι στο μέλλον θύμα ε, βίας λόγω φύλου. Γι' αυτό ζητούμε μια στρατηγική στήριξης και σεβασμού. Επίσης ε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι διάκρισης, η υποχρεωτική έκτρωση, η αποκλεισμό από το δικαίωμα στη μητρότητα ή στην υιοθεσία αυτή και αν είναι διάκριση. Είναι πραγματικά απάνθρωπη μεταχείριση μερικέ φορέ των γυναικών με αναπηρίε. Θέλουμε και δείκτε για να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση αυτών των γυναικών. Δείκτε με βάση το φύλλο, με βάση την αναπηρία, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Αναπηρίες και να καλύπτονται και όλοι οι τομεί. Επίση, το άρθρο 5 των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μιλούσε για τη χειραφέτηση των γυναικών, την ενδυνάμωση των γυναικών, των γυναικών με αναπηρίες. Μόνο έτσι θα δώσουμε ε, δύναμη και στην ανθρωπότητα. Σήμερα έχουμε ευκαιρία για να μάθουμε, να νιώσουμε, να διδαχθούμε και να δημιουργήσουμε. Κάποια γυναίκα με αναπηρία μου είπε ε, χαίρομαι που είμαι γυναίκα. Έχω μία αναπηρία, αλλά έχω και πάρα πολλέ ικανότητε, όπω και οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μου. Και είμαι κυρίω άνθρωπο, με όλα τα δικαιώματα που έχω. Και ελπίζω ποτέ να μην πρέπει να δικαιολογήσω γιατί το δικαιώμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Δεστάρα Φεραγκούτ Η Επίτροπο θα Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε κυρίε και κύριοι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ανάπτυξη για όλους, η ισότιμη αντιμετώπιση είναι στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μείνει κανείς αποκλεισμένος. Ευχαριστώ την κυρία Σταράς Φεραγούτ, την Επιτροπή των Γυναικών που προβάλλουν το θέμα αυτό, το θέμα των γυναικών δηλαδή με αναπηρίες. Η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρίες στην κοινωνία και να προαγάγουν την ισότητα των φύλων. Δύο παραδείγματα. Ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας για την οποία έχουν, κλείσει, έχουν καταλήξει νομοθέτες σε μια προσωρινή συμφωνία που ε, εξασφαλίζει σημαντικέ αλλαγέ για κύρια προϊόντα και ε, Υπηρεσίε και ταυτόχρονα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα. Ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να δώσουμε υποστήριξη σε εκείνους που μεριμνούν για άλλου μέλη τη οικογένεια, του κυρίω γυναίκε, για να μπορούν να συνδυάσουν και τον οικογενειακό βίο και βίο προσφορά στους άλλου, αλλά και τον επαγγελματικό. Και αυτό νομίζω θα επιτρέψει να εξισορροπηθούν οι ανάγκες ε, και πιστεύω ότι θα κλείσει σύντομο ο τριμερής διάλογο για τα τρία συγκεκριμένα ζητήματα που θέτεται. Μαζί με όλα τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Αναπηρίες αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη στήριξη της πορείας ε, εφαρμογής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σύμβασης προς, το, προς τον ορίζοντα του 2020 και αποτελεί κομμάτι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη δημιουργία ευφύους Βιώσιμη ανοιχτή σε όλου ανάπτυξη, η κοινωνική συμμετοχή, η δυνατότητα συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία είναι εκτρόνου κανένα φόρο όρος για την επιτυχία τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή αξιολογεί την υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγικής Αναπηριών, αξιολόγηση η οποία θα καλύψει κάθε επιτυχία αναπηρία, κάθε είδο αναπηρία και ιδιαίτερα θα δώσει έμφαση στην κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με την διάκριση λόγω φύλου των ατόμων με αναπηρίες και οπωσδήποτε θα κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε στο δυνατόν περισσότερους παράγοντες στην διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπωσδήποτε με βάση άλλωστε και το ψήφισμα του 2017 που περιλαμβάνει και τις ε, παρατηρήσει Επιτροπής των Γυναικών για ολοκληρωμένα δεδομένα, αξιόπιστα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας πολιτικής επιλογής και γραμμής. Ήδη έχουμε κατανομία φύλλο ανα, αναπηρία των δεδομένων μας, ε, όπως τα συλλέγουμε εν ώψη της χάραξης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεδομένα τα οποία αποτελούν μια αντικειμενική βάση για τον εντοπισμό διακρίσεων που οφείλονται στο φύλλο Επί παραδείγματι έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις ε, κινδύνου φτώχειας ή ανεργίας πολύ, μεγάλη, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες με αναπηρία. Στον τομέα όμως της εκπαίδευσης σημειώνουμε ότι είναι πολύ ψηλότερο το επίπεδο των αγοριών με αναπηρίες που εγκαταλείπουν το σχολείο παρά των κοριτσιών με αναπηρίες βεβαίως. Η ισότητα των φύλων ε, είναι μια διάσταση που προβάλλουμε και στις εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς και τονίζουμε στις χώρες εταίρους ότι πρέπει να βελτιώσουν την ε, μέθοδο συλλογής δεδομένων και μάλιστα την κατανομή αναφύλων και ε, αναπηρίες ε, και έτσι να υπάρχει μια πλήρης ανάλυση δεδομένων για κάθε έργο ή πρόγραμμα που μπορεί να αναπτύσσεται σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Θα ήθελα επιτέλου να αναφερθώ στα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή ηθελα επιτελου να αναφερθω στο οσα κανει η ευρωπαικη επιτροπη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Εκλογικό Γίγνεσθε. Η συνάδελφος Γιώροβα έχει εκδώσει δήλωση για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωεκλογές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ολομέλεια της 5ης Ιουλίου του 2018. Όπως ε, σημείωσε λοιπόν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Γεωρούβα, η σύσταση της Επιτροπή του Φεβρουαρίου του 2018 αναφέρεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στόχο έχει την προαγωγή της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε ε, για όλους και κυρίως ε, για τα άτομα με αναπηρία. Ε, για εφέτος έχουμε ε, προβλέψει μια ειδική ε, συνεδρία γι' αυτό, συμμετοχή δηλαδή ατόμων με αναπηρίες και προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν στο εκλογικό γίγνεσθε. 26 και 27 Νοεμβρίου συγκεκριμένα την εβδομάδα την τρέχουσα έχουμε αφιερώσει ένα συνέδριο για τα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στο θέμα της προαγωγής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και μια ανοιχτή προς όλους δημοκρατική κοινωνία. Τέλος. Θα ήθελα να φέρω ότι η οδηγία για την προσβασιμότητα των φορέων ε, του δημοσίου και ο σχετικός ιστότοπος που έτεθησε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2018 αποτελεί μια βάση ενημέρωσης για τους ε, φορείς του δημοσίου των κρατών μελών και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Τάισεν και τώρα το λόγο έχει για ένα μισή λεπτό η κυρία Κοσλόφσκα ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη Ρόζα Εστέρας για το αρτιότατο ψήφισμά τη με θέμα τη γυναίκε με αναπηρίε. Στην Ευρώπη διαβιούν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίε, 46 εκατομμύρια είναι γυναίκε. Μόνο 18% από τι γυναίκε αυτέ έχουν κάποια θέση απασχόληση. Και κυρίως οι γυναίκες ασχολούνται και φροντίζουν άτομα με αναπηρίες. 80% αυτών εργάζονται ατύπως και αμυστοί. Πρόκειται για τον κλειστό κύκλο των ανισοτήτων, των ατέρμονων προσπαθειών και της αδικίας. Γιατί τόσο λίγες γυναίκες ε, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. Τι διατάξει, η έλλειψη διατάξεων δημιουργούν προσκόμματα στην οικονομική ανεξαρτητοποίηση των γυναικών με αναπηρίε. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, δεν είναι θέμα μόνο αναξιοποιητών ταλέντων και ικανοτήτων. Είναι και θέμα ανθρώπινη αξιοπρέπεια που συνδέεται με την ανεξαρτησία και την πλήρη συμμετοχή στον κοινωνικό και οικονομικό βίο. Άλλωστε, οι σημερινέ τεχνολογίε, όπω λέει και το ψήφισμα, δίνουν στους, στα άτομα με αναπηρίε ασύγκριτα περισσότερε δυνατότητε από παλιά για φυσιολογικό βίο και αυτοεκπλήρωση. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να εφαρμόσουμε τη συμβάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίε και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τι Αναπηρίε. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν και να εφαρμόσουν πλήρω τι διατάξει για τα άτομα με αναπηρίε. Και επίση θα πρέπει να, συμπεριλάβουν τι διατάξει οικονομικού σχεδιασμού, την αξιοποίηση των ψηφιακών ε, τεχνολογιών και τη ιατρική προόδου, ώστε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία, την προσληψιμότητα και την αίσθηση δικαιοσύνη των ανδρών και γυναικών ατόμων Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Κοσλόφ Σκαράγεβιτ. Το λόγο έχει η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, ατόμων ε, και των γυναικών με αναπηρία, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για το θέμα αυτό. σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει καθημερινά να συζητάμε με τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Όταν μιλάμε για τον, ευρωπαϊκό, τον κοινωνικό πυλώνα, δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να μειώσουμε και να εξαλείψουμε την διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή σε ό,τι αφορά τους μισθούς κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για φτώχεια, για κοινωνικό αποκλεισμό. Οι γυναίκες με αναπηρία δεν μπορούν να συνεμετανασχολούν στην αγορά εργασία. Δεν μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή και προφανώς η εργασία αποτελεί πηγή εισοδήματο, αλλά και ευκαιρία α, να έρθει κανείς σε επαφή με άλλα άτομα. Τίφερε το θέμα και των συντάξεων για τις γυναίκες με αναπηρία. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με αναπηρία. Και δεν μπορούμε κατά συνέπεια να επιλύσουμε το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης στη σωστή του διάσταση. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει εφαρμοστική διάταξη από τα ταμεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα έχουμε την κυρία Βυσνιέσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Η ευαισθησία μας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες φαίνεται και με την εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των ατόμων της αναπηρίας. Αυτό όμως είναι κάπως υποκριτικό γιατί ε, τώρα που πλησιάζει η Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με Αναπηρίες ε, αρχίσαμε και στο Κοινοβούλιο να μιλούμε για τα θέματα αυτά ε, των ατόμων με αναπηρίες που θα πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες και δυνατότητα για παιδεία, για επαγγελματική σταδιοδρομία, για πρόσβαση σε καλό πολιτισμό. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας για να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά εδώ όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μείνει σύσσωμο και πέραν των ε, κομματικών διαφορών θα πρέπει να αναλάβουμε δράσεις που να επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να ζουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Και κρίμα που στο ψήφισμα αυτό και κοιτάω προς την αριστερή πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβάνεται και θέματα ισότητας φύλων. Ε, νομίζω ότι η αλλαγή φύλου. Ευχαριστώ, κύριε Βυσνέσκα. Η κυρία Μέτσε έχει το λόγο, αλλά πού βρίσκεστε, άλλαξατε θέση. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σεβαζόμαστε πραγματικά την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Όχι, γιατί άνθρωποι με αναπηρία εξακολουθούν να βρίσκονται σε διακριτική, σε μειονεκτική θέση και κυρίως οι γυναίκες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την εργασία αλλά και την προσωπική και ε, ανάπτυξη. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ευτυχία, όλοι έχουν δικαίωμα να ε, καθορίζουν τη ζωή τους. Μια ζωή όπου η σεξουαλικότητα δεν αποτελεί ταμπού, όπου μπορεί κανείς να ασκήσει ελεύθερα την σεξουαλικότητά του και που το όχι σημαίνει όχι, που έχει δικαίωμα να ιδρύσει μια, να δημιουργήσει οικογένεια, να παντρευτεί, να ζήσει μαζί με τον ή την σύντροφό του. Και ακριβώς λοιπόν στους τομείς αυτούς οι γυναίκες ε, που έχουν αναπηρία χρειάζονται την υποστήριξή μας και την καθοδήγησή μας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται για συμπόνια. Μιλάμε για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μέτς. Για ένα λεπτό, ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποποιείται των ευθυνών τη, γιατί έχει επιδεινωθεί η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίε, κυρίω των γυναικών, που υφίστανται διπλέ διακρίσει. Οι πολιτικέ λιτότητε που προωθεί συρρυκνώνουν τα οικονομικά και επαγγελματικά εργασιακά δικαιώματα και ε, ε, Δυστυχώ περιορίζονται και οι εθνικέ επενδύσει στην παιδεία, στην υγεία, κάτι που επηρεάζει αυτή την κοινωνική επιδείνωση των ατόμων με αναπηρία ε, στερούνται μερικέ φορέ και στοιχειωδών θεμελιωδών δικαιωμάτων οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν δικαιώματα πολλέ φορέ στην αγορά εργασία, δεν έχουν καλή πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, ε, είναι μονίμω καταδικασμένοι στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, στην ελληπή κοινωνική προστασία, δεν έχουν μέσα βιοποριστικά, δεν έχουν καλή πρόσβαση στη, στη δημόσια παιδεία, δεν, μπο, δεν, χαίρουν των προϋποθε, δεν που έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Επίση δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη τροφαρμακευτική περίθαλψη. Ε, υφίστανται περιορισμού στην κινητικότητα, δεν έχουν καλή πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό μεταξύ άλλων. Γιατί οι δημόσιες πολιτικές δεν δίνουν απάντηση δυστυχώ στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόιντρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τι γυναίκε με αναπηρία στην εκπαίδευση, την ε, εργασιακή ζωή στον, στον τομέα της υγείας θα πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο παρά το γεγονός ότι δεν συμβαίνει αυτό σε πολλούς ε, τομείς. Οι γυναίκες ε, με αναπηρία συχνά έχουν ζήτημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά και την πρόσβαση και σε άλλους τομείς και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με βία θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την κατάσταση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το κείμενο αυτό. Επιστούμε την προσοχή στα προβλήματα των γυναικών με αναπηρία και ελπίζω ότι για τα κράτη-μέλη αυτό θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να εξασφαλίσουν υπηρεσίες καλύτερη ποιότητα. Ωστόσο, να διευκρινίσω ότι υπάρχουν ζητήματα θέματα τα οποία, τα οποία διαφωνώ σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την παρατρύνση για την έγκριση της συμφωνίας της ε, Κωνσταντινούπολης, σε ό,τι αφορά τη βία και την υγεία των ε, γενικών ατόμων. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζουν αυτά στο κείμενο και δεν τα υποστηρίξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει κ. Μπενιφέκ. Δεν είναι εδώ. Διαδικασία Κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά μέσα από τη συζήτηση για τις διακρίσεις των γυναικών των ατόμων εκείνων που έχουν αναπηρίες αναδεικνύεται ένα μείζον θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι οι γυναίκες που έχουν προβλήματα αναπηριών δεν τη χάνουν μόνο τι δυσμενού διακρίσεως αλλά η δυσμενή διάκριση υφίσταται σε όλο το φάσμα των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είναι πρωτοπόρο και πρωταγωνιστή να εφαρμόζει πλήρω και απόλυτα την αρχή ότι δεν πρέπει να υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και παραμένει μια βασική και ατράνταχτη απαραβίαστη αρχή που οφείλουν όλοι να εφαρμόζουν και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε μόνο με λόγια και διακηρύξεις. οι διακηρύξεις είναι εδώ και υπάρχει σήμερα η δυνατότητα η ευρωπαία η ευρωπαϊκή επιτροπή να δεσμευτούν ότι θα υπάρξει πλήρης και απόλυτη εφαρμογή στην ισότητα των φύλων και θα επιβληθούν κυρώσεις σε όσα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την ισότητα των δύο φύλων. μόνο έτσι θα γίνει πράξη η εφαρμογή πλήρης και απόλυτη του σεβασμού της ισότητας των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ κύριε Χριστοφόρου. Stevens. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ζητά προσοχή με το κείμενο αυτό για το θέμα των γυναικών με αναπηρία. Οι γυναίκες με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν ζητήματα διαφυλικής, διακριτικής μεταχείρισης λόγω του φίλου του και λόγω τη αναπηρία του. έχουν πολύ περισσότερε πιθανότητε να γίνουν θύματα σεξουαλική βία σε σχέση με γυναίκε που δεν έχουν αναπηρία και επίσης υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και στην πολιτική και γι' αυτό λοιπόν πολλές γυναίκες με αναπηρία θεωρούν και αισθάνονται απομονωμένες στην κοινωνία. Ελπίζω η Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων να προωθήσει την στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων το 2030 προκειμένου η διακριτική μεταχείριση για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία να αντιμετωπιστεί με σοβαρό τρόπο. Η ισότητα και ο σεβασμός των ε, γυναικών με αναπηρία. Δεν θέλουμε άλλα λόγια, θέλουμε πράξεις και τώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Στίβενς και στο τέλος ε, ο κύριος Μαγιάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει αποκαλύψει ότι πραγματικά υπάρχουν δυστυχώς διακρίσεις κατά των γυναικών οι οποίες είναι άτομα με αναπηρία. Και αυτό που χρειάζεται είναι να μην λέμε πολλά λόγια να μην βρίσκουμε αφορμή ότι στις 3 Δεκεμβρίου θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία και κάνουμε επευκαιρία αυτή τη συζήτηση. Διότι εδώ πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και το έχουμε πει επανειλημμένα σε παρεμβάσεις μας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πρέπει να εφαρμοστεί η σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις διακρίσεις κατά των γυναικών οι οποίες είναι αμαία και αυτό το βλέπουμε διότι υπάρχει δυσκολία στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. πολύ δε περισσότερο στην ελλάδα όπου εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες διακρίσεις και λόγω των μνημονίων έχουν μειωθεί και τα επιδόματα τα αναπηρικά. επομένως χρειάζονται μέτρα συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση με την παρέμβαση της Επιτρόπου κ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Η συζήτηση αυτή έδειξε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι η στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση που επιλέξαμε και για την ισότητα των φύλων αλλά και για τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες. Η ισότητα των φύλων, οι ίσες ευκαιρίες και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας ε, είναι σημαντικές αρχές ε, του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το διακηρύξαμε πανηγυρικά πριν από μία περίπου χρονιά όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και σίγουρα ε, η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια θα συμπεριληφθεί στη, στον προβληματισμό για τη μορφή και το περιεχόμενο που θα έχουν στο μέλλον οι πολιτικές ε, για τις αναπηρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των ε, ε, οργανώσεων που τους αντιπροσωπεύουν σε όλη αυτή τη σκέψη. Και φυσικά προσβλέπω στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών μελών και θέλω να γίνουν ισχυροί σύμμαχοί μας προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή και έμπρακτη εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Τάισεν και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και στο τέλο τη συζήτηση ε, έχουμε το ψήφιμα σφίσμα V8 520 του 2018 και η ψηφοφορία επ' αυτού θα λάβει χώρα σήμερα. Διακόπτεται η Σύνοδος μέχρι την έναρξη των ψηφοφοριών.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

Christine, Christine. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε. Αν θέλουμε να τελειώσουμε εγκαίρως, Λοιπόν, όσο κάθεστε, να σας ενημερώσω ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μία αντιπροσωπεία από το Μαζλισί Ολί με επικεφαλή στο Σαρίφ Ζοντά. Η αντιπροσωπεία είναι εδώ στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην 7η Επιτροπή Διακυβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τατζικιστάν. Είμαστε ε, ιδιαίτερα ευτυχείς που θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη συνάντηση που θα ενισχύσει τις σχέσεις και τη συνεργασία μας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό δείχνει την κοινή μας δέσμευση για τα δημοκρατικά δικαιώματα, τον ε, πολιτικό πλουραλισμό μέσω του κράτους δικαίου από πλευρά ολοκλήρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, σας ε, εύχομαι επιτυχή συνεδρίαση και μια ευχάριστη παραμονή στην Ευρώπη. Θα, θα επιληθεί το θέμα που αναφέρετε κύριε. Σας είδα κύριε, σας είδα κύριε. Αλλά πρώτα είδα την κυρία. Ωραία, ωραία. Ρυθμίστηκε το θέμα αυτό. Κυρία Ward, έχετε κάποιο πρόβλημα διερμηνίας. Όχι. Madame Κυρία Ward. Συνάδελφοι, στα πλαίσια της ε, σημερινής ε, ιστορικής ε, ομιλίας για, από δύο νομπελίστες εμείς που κερδίσαμε το Νόμπελ το 2012 θέλω να σε ενημερώσω ότι χθες στις 28 Νοεμβρίου ήταν η 7η επέτειος της δήλωσης ε, των Βρυξελών που είναι μια διακήρυξη για την ειρήνη που υπεγράφει εδώ στο σώμα μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την αιγίδα του Τζιάννη Πιτέλα που ήταν ε, αντιπρόεδρος. Αυτή η δέσμευση ενθαρρύνει προγράμματα και δράσεις που προωθούν την ειρήνη με την πιο πανανθρώπινη έννοιά της με τη σημασία που έχει για κάθε άτομο. Βασίζεται στις πανανθρώπινες ιδέες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης που αναφέρονται στο προήμιο της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώθηκαν από την Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. Οπότε, ας θυμηθούμε, συνάδελφοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πάντα θα είναι ένα εγχείρημα που προωθεί την ειρήνη. Πρόεδρος, να περάσουμε στις ψηφοφορίες απευθείας με την έκθεση Dalton για την εφαρμογή του σταδίου Ευρώ 5 για την έγκριση του τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων και τετρακύκλων. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Έχετε καθίσει όλοι. Ε, τότε πέρας. Εγκρίνεται. Περάσουμε στην έκθεση Γκέριγκερ, The Udenberg Πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνατών που είναι, να, να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση τιμωρία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέραμε τώρα στην έκθεση Ντάλι εκ νέου δέσμευση των υπολείπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προ στήριξη τη εφαρμογή των αποφάσεων για να εφαρμοστούν οι αποφάσει του Συμβουλίου. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Η κυρία Νταλή ήθελε να πάρει το λόγο. Θα είναι πολύ σύντομο, μην ανησυχείτε. Η κυρία Νταλή. Ευχαριστώ. Με βάση του άρθρου 95.4 το θέμα αυτό θα πρέπει να επανέλθει στην Επιτροπή για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Ωραία, να ψηφίσουμε την πρόταση της ηγήτριας κατά αποχές δεκτό. Θα επανέλθει στην αρμόδια Επιτροπή. Έκθεση David Martin. Προσχώρηση τη ΑΜΟΑ στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών του Ειρηνικού. Πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην έκθεση Γουαλτιέρη. Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μυστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Η υποψηφιότητα του κυρίου Ανδρέα Αέρια επικυρώνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση τη κυρία Γουαρδεδιαβάλ Ρούμπιελ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Τμήματο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Για το EL ε Attica Publishing. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Με την αναγκαία πλειοψηφία. Έχουμε την έκθεση Φαγιόν για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Έχουμε μια σειρά τρόπολογίες από την αρμόδια επιτροπή, τις οποίες θα ψηφίσουμε από κοινού υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές Θα ελέγξουμε αυτή την πρώτη ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Δεκτές. Τροπολογία 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 9 ε, ναι, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 40 υπέρ. Α, καλά, να ελέγξουμε τη 13. Ελέγχουμε, άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται πέρας Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 21 ντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Λοιπόν, η 51 καταπίπτει, περάμε στις τροπολογίες 22D και 52D υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτές 23 ε, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 54 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Το 26 ονομαστική. Άρχισε. Πέρας. Δεκτή. Οπότε 56 σε 1 υπέρ, σε 2 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 CP3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 ντε και 57 ντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 56 CP4 η επόμενη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε την 56 CP5 την επόμενη υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Αμφίροποι. Ελέγχουμε. Την 30. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 59 αντί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε καλά την 31 την 31 μάλιστα ελέγχουμε την 31 πέρασε Δεκτή. Λοιπόν, η επόμενη καταπίπτη... Α, όχι. Ψηφίζουμε. 56 CP6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Εδώ έχει ζητηθεί ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 60. Υπέρ. 60 CP3. 60 CP3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 35 άρχεται πέρας δεκτή 61 CP1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38D υπέρ κατά αποχές ελέγξουμε. 38D. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική 64. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε τη 44 με ονομαστική επίσης. Άρχεται. Ψηφίζουμε ονομαστική 44. Πέρας. Δεκτή. 45 και 66 από κοινού άρχεται. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη, υπέρ, υπέρ καλύτερα. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, ξέχασα, ξέχασα. Πήδηξα την 68. Θα ήταν κρίμα. 68 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ονομαστική επί της 3. Άρχεται. Επί της 3. Πέρας. Δεκτή. Ονομαστική επίση ε, για την 5 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Ονομαστική και για την 6 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Ονομαστική επί της 7 άρχεται. Τώρα άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 12 επίση ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 15 ονομαστική άρχεται. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Να ψηφίσουμε την 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. Γιατί είναι αμφιερωπή. 14. Πέρας. Δεκτή. Οπότε ψηφίζουμε τη 15. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Και ψηφίζουμε τώρα την τελική ψηφοφορία, πρόταση της Επιτροπής Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Κυρία Φαγιόν, ε, να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ το θέμα να επανέλθει στην Επιτροπή για να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τον κανόνα 59.4. Ευχαριστώ Το άρθρο 59.4 του κανονισμού. Πρόεδρος. Ωραία. Ψηφίζουμε την πρόταση της συγγήτριας υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Άρα πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την πρόταση αυτή της συγγήτριας. Πέρας. Δεκτή. Θα επανέλθει στην Επιτροπή. Λοιπόν, ε, δεν θα πούμε συγχαρητήρια. Έκθεση τα Παρντέλ κοινή κανόνε εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών. Ονομαστική επί της τροπολογίας 3. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρούται με αυτόν τον τρόπο. Περνάμε στην αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού. Διχρωμικό νάτριο. Ποιοι είναι υπέρ του ψηφίσματος. Ποιοι είναι κατά. Αποχές παρακαλώ. Δεκτό. Περνάμε στο θέμα το σκάνδαλο Καμέξ οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Τροπολογία 46. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 λοιπόν υπέρ. Παρακαλώ, ε, να σηκώνω τα χέρια, δεν βλέπω τίποτα. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά, Αποχές. Αφού δεν βλέπω τίποτα θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την 4. Πέρας. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ονομαστική για την 6. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Ονομαστική επίσης για την 16. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 17 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21-48-71 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε, άρχεται, ελέγχουμε τις 21-48-71. Πέρας. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τις 22 και 72. Από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Ελέγχουμε την 49. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 και 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52-75 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Μ, αμφίβολο. Ψηφίζουμε, ελέγχουμε 52 και 75. Άρχεται. Πέρας. Δεκτές. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ θέλετε να ελέγξουμε την 53 μα κανείς δεν σήκωσε χέρι του μπας περιπτώσει ωραία ελέγχουμε την 53 άρχεται πέρας δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική για την 26 άρχεται πέρας δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30, 55 και 77 έχουν αποσυρθεί οπότε ψηφίζουμε την 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Η παράγραφος 10. Το αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31, 57, 79. Μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ονομαστική για τις 58 και 80. Θέλετε να ελέγξουμε. Α, θέλετε να ελέγξουμε την προηγούμενη. 31 επανερχόμεθα. 31, 57 και 79 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε ονομαστικά για την 58 και την 80. Άρχεται. Πέρας. Δεκτές. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ονομαστική για την 34. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ορμαστική επίσης για την 35. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Ψηφίζουμε 36 και 61 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 60 και 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές έχω αμφιβολία να ελέγξουμε 84 πέρας εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8, 42, 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 9, 43, 65 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Ονομαστική για το 2D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 10 Ανατασχυρώσει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική για την 11. Άρχεται η ψηφοφορία. 11. Πέρας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 66. Ανάτες χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι βέβαια. Ψηφίζουμε. Για έλεγχο. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την 12. Άρχεται ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1368 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1469 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 15 ονομαστική ψηφοφορία. Έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το ρόλο τη Γερμανική Υπηρεσία Κοινωνική Μέρημνα Παιδών και Νέων, Jugendamt, τι δεξιωριακέ οικογενειακέ διαφορέ. Ξεκινάμε με την ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 5, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Πρώτο τμήμα. Αρχικό κείμενο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Να έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ανάταση χειρός 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία 8D. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφο 9, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε 23. 23 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφο 9, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ε, για το πρώτο τμήμα, άρχεται αυτή. Πέρα. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, άρχεται αυτή. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπεται. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11, αρχικό κείμενο, 3 τμήματα, πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13, ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία αρχικό κείμενο, παράγραφος 14, πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, ανάταση χειρός, 12, 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το 13D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 διανάταση χειρό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν είναι και πολύ σαφέ να ε, επαληθεύσουμε. Τροπολογία 14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε και το 15. Πέρας. Απορρίπτεται. Δυνατές ισχυρός 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για να επαληθεύσουμε για την 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πράγματι. Αρχικό κείμενο, παραγράφος 22, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Άρχεται αυτή. Με συγχωρείτε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι αμέσως. Τώρα. Εγκρίνεται. Δυνατή ισχυρό 20. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, δεν είμαι βέβαια. Να ψηφίσουμε για την 20. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, η αναφορά 13 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές. Δεύτερο τμήμα της 13. Υπέρ, ε, συγγνώμη, Πέρας. Ήταν πραγματικά πολύ κοντά η ισοψηφία ε, εγκρίνεται. Επειδή είναι αρχικό κείμενο, σε, σε περίπτωση ισοψηφία, εγκρίνεται το κείμενο, συνάδελφοί μου. Ήταν πολύ αβεβαιό όμω το τι συμβαίνει. Αιτιολογικέ σκέψει, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ξανά, ε, ξανά είναι ασαφέ. Ψηφίζουμε για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική ε, σκέψη σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπήρχε και τέταρτο τμήμα. Ε, ονομαστική ψηφορία πάλι. Άρα δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δυνάτες ισχυρός 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, αρχικό κείμενο, διατμήμα το πρώτο τμήμα, ε, σε ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. δεν κρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Έρχεται αυτή. Αιτιολογική σκέψη ε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη F. Άρχεται αυτή. Πέρας. εγκρίνεται. Δυνατές ισχυρό 17 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Έλεγχο. τροπολογία 17, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την 3D. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρα. Εγκρίθηκε. Κυρία Βίξτρομ, έχετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα διαδικαστικό. Συνάδελφοι, θα ήθελα το όνομά μου να διαγραφεί από το ψήφισμα αυτό της Επιτροπής Αναφορών για την Jugendamt, διότι το κείμενο που μόλις ψηφίσαμε δεν είναι το σχέδιο κειμένου που πρότεινα εγώ. Ε, τροποποιήθηκε και αλλοιώθηκε από τις προφορίες στην Επιτροπή μας ε, και μάλιστα επί της ουσίας γι' αυτό το όνομά μου θέλω να διαγραφεί εντελώς από τη σύνταξη του κειμένου. Δεν είναι το δικό μου το κείμενο και δεν θέλω τέτοιο να παραμείνει στα, αρχικά, στα πρακτικά. Πολύ ωραία, καταγράφουμε το έτοιμά σας, κυρία Βίξτρομ. Περνάμε στην έκθεση των κυρίων Λάγκε και Ρούμπιχ για τον ΠΟΕ πορεία προς το μέλλον. Ε, ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίθηκε. Έκθεση Μακάλιστα. Έκθεση του 2018 για τη Σερβία. Παράγραφος 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 και 3 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Καθόλου. Ε, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 4 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Σαρδάμ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την έκθεση Σόλτε, έκθεση το 2018 για το κοσυφοπαίδιο. Παρά αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. σε ισχυρό πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δύο Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν είναι σαφέ να επαληθεύσουμε για τη δεύτερη τροπολογία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παραγραφό 12 αρχικό κείμενο άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 42 τα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βάγκλ. Ε, έκθεση το 2018 για την πρώην Γεκλουσαυκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Διανάταση ισχυρός, τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρώτη και δεύτερη τροπολογία από κοινού. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνονται. 14. Μην ο κύριος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Μονομαστική ψηφοφορία για την 5. Άρχεται, αυτή, η ψηφοφορία. 5. Πέρας. Εγκρίνονται. Διανάτες ισχυρός 4. Υπέρ. Κατά. Κανείς δεν λέει τίποτα. Υπέρ. 4. Να. Επιτέλους. Ε, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παραγραφούς 55-7 ναι, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές Αμφιβάλλω λίγο για το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για να ελέγξουμε. 6. Επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα για την ατολική σκέψη Α. Διένατε ισχυρό υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο και αιτιολογική σκέψη F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα νομιστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Χωρίς διακοπέ, περνάμε στην έκθεση Φλέκενστάιν, έκθεση του 2018 και την Αλβανία. Παράγραφος 1. Διανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. αποχές Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε προφορική τροπολογία σε αυτή τη φάση, παρακαλώ. Yeah, ναι. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μια προφορική τροπολογία 21α. Σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και οι Ρωμά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αναπαραγωγικής υγείας και δεν γνωρίζουν την διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών. Ζητάει λοιπόν από τις αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν καλύτερη πληροφόρηση για αυτές τις υπηρεσίες και να φροντίσουν να είναι προσβάσιμες ε, και από πλευράς τιμών. Υπάρχει αντίρρηση για την τροπολογία αυτή. Αν θέλετε ε, να προβάλλετε αντίρρηση, ε, δεν βλέπω 40 άτομα. Προφορική τροπολογία ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά,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 6D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. 4 ψηφίζουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται. 7D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. αντί Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Να γκρίνεται. Και τώρα η έκθεση του κυρίου Καν. Η προάσπιση τη ακαδημαϊκής ελευθερία στην τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρώτο τμήμα για την τοπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε αυτή. εγκρίνεται. λογική αναφορά 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ε, πρώτη, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ε, άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, πρώτο, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, ε, ε J, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, λογική σκέψη L, υπέρ, Κατά αποχέ εγκρίνεται. λέξη σκέψη. Εν. Αρχικό κείμενο διατμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Κατάσταση των γυναικών με αναπηρίε. Πρόταση ψηφίσματο τη Επιτροπή για Δικαιώματα των Γυναικών και τη Ισότητα των Φύλων. Αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο, ε, ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Η άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11, 4 τμήματα, πρώτο τμήμα. Δυνατέ ισχυρό υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, αρκετά αυτή. Και πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, αρκετά αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 19, πρώτο τμήμα, διάνατος ισχυρός υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Διένατας ισχυρός 20. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 24. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 26 υπέρ. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αμφιβάλλω λίγο. Οπότε 26 έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παραγωγό 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 35. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 37. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία μάλλον. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 45. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφορία. Άρχεται αυτή. 45. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την τροπολογία σε 2. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Μπορεί να ψηφίσει. Ναι, ε, τελείωσε. Εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη G σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη H, πρώτη σε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε αιτιολογική σκέψη L, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ναι, και εγώ αυτό θα Έπρεπε Να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Ζητούμε συγγνώμη από το Προεδρείο. Ξαναπάμε πίσω στην αιτιολογική σκέψη H. Έπρεπε να έχουμε ψηφίσει το αρχικό κείμενο. Οπότε ψηφίζουμε αυτό το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρέπτει. Εντάξει λοιπόν, αφού θέλετε να ελέγξουμε, να παληθεύουμε για το αρχικό κείμενο της εντολεξίευσης H, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. Εν... η σκέψη M. Ονομαστική ψηφορία άρχεται αυτή. Ναι, ας ε, ανοίξουμε και τα μηχανήματα. Ε, πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το τροπολογία 4. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική, ε, μάλλον συγγνώμη, τροπολογία 5. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Γιατί σκέψη Β, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρα. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Thank you so much. Oké, okay, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégák! Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Λοιπόν, αν πρέπει να φύγετε από την αίθουσα παρακαλώ διαλυθείτε ησύχως για να ξεκινήσουν οι ομιλητές.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 να σας ενημερώσω ότι λόγω των πολλών επεξηγήσεων ψήφου πρέπει να διακόψουμε το αργότερο στις 1.30 Συνάδελφοι, παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα ήσυχα Λοιπόν, κάποιοι ομιλητέ δεν θα λάβουν τον λόγο. Όσοι δεν μιλήσουν, παρακαλώ να υποβάλουν εξηγήσει ψηφού γραπτός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο ψήφισμα είναι το σκάνδαλο και τα παραθυράκια στο νομικό πλαίσιο. Ο κ. και έχει τον λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό με το ψήφισμα αυτό είναι ακριβώς να κατονομάσουμε την χώρα που έκανε όλα αυτά τα σκάνδαλα και είναι λυπηρό ότι η Γερμανία ε, μια τόσο σημαντική χώρα έχει τόσα πολλά παραθυράκια στο νομικό της σύστημα ώστε μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα μιλάμε για απόλυες σε φόρους 55 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ σε 11 ε, κράτη-μέλη επειδή ήταν κάποιοι δικηγόροι και τραπεζίτες ανέντιμοι. Τα λεφτά αυτά μπορούσαν να έχουν πάει στο γερμανικό στρατό, παραδείγματος χάρη, και να τον χρηματοδοτήσουν πλήρως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε το νομικό μας σύστημα για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και να κάνουμε αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Ροζάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακοβέ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκάνδαλο αυτό μας έδειξε και πάλι ότι όταν οι αρχές κάνουν τα στραβά μάτια οι δημοσιογράφοι κάνουν τις έρευνες και αποκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτοί αποκάλυψαν πως 55 δισεκατομμύρια ευρώ απεκρέβησαν από έντιμους ανθρώπους, ε, από τους έντιμους φορολογούμενους και χρειάστηκαν 10 χρόνια για να αλλάξει η Γερμανία την νομοθεσία ε, περί μερισμάτων. Η Γαλλία, η Δανία και η Ολλανδία επίσης έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά οι αρχές ε, σκοντάφτουν σε ζητήματα διαδικαστικά γραφειοκρατίας ε, και το αποτέλεσμα στην πράξη είναι ότι κάποιοι κλέβουν και μένουν ατιμόρυτοι. Το ΚΑΜΕΞ είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη κομπίνα στην ιστορία της Ευρώπης και αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε μια γρήγορη ευρωπαϊκή απάντηση χτες, όπως λέμε, για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Σας ευχαριστώ. Για το ECR, συνάδελφος Ρούνεν Λέρνερ. Σας ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχασαν λόγο κομπίνας με τα μερίσματα τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Το φορολογικό αυτό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε χάρη σε κάποιους δημοσιογράφους. Και πάλι έχουμε μια κατάσταση όπου οι αρχές δεν ε, διέδωσαν τις πληροφορίες για το σκάνδαλο αυτό. Και αυτό ακριβώς περιγράφει το πρόβλημα του να μπαίνουν βγαίνουν από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κάποιοι παραδείγματο χάρη είναι ένας φορολογικός σύμβουλος μετά απασχολήθηκε από τον τραπεζικό τομέα για να αναπτύξει αυτά τα κόλπα και σύμφωνα με τις πηγές ε, ήταν κάτι το νόμιμο είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πώς ε, λειτουργούν τα συστήματα και πώς έπαιρναν ε, άνθρωποι επιστροφή φόρου χωρίς να έχουν πληρώσει φόρο το σκάνδαλο αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και ο επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Ε, με χαρά μου υπερψήφισα. Σα ευχαριστώ. Κύριο Σανκέλη έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φορολογική αυτή απάτη, όπως αναφέρθηκε, κοστίζει, κόστισε στα κράτη-μέλη γύρω στα 55 δισεκατομμύρια. Τεράστια ποσά μέσω πολύπλοκων συμφωνιών που δεν εξυπηρετούσαν κανένα σκοπό παρά μόνο το να εισπράττουν ε, επιστροφή φόρου χωρίς να έχουν πληρώσει φόρο. Λιστεύτηκαν έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση φορολογικής απάτης, αλλά το σκάνδαλο αυτό μας δείχνει πως υπάρχει ένα κενό στην εφαρμογή, την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Λογικό είναι να έχει προκαλέσει οργή το σκάνδαλο αυτό και απαιτείται δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτή η φορολογική κλίμακα μεγάλης, αυτή η φορολογική απάτη μεγάλη κλίμακα πρέπει να κατασταλεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριο Χάναν. κύριε Αντιπρόεδρε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το σύστημα δούλεψε. Οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους και η νομοθεσία άλλαξε. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι υπόλοιποι τώρα πετάμε κι εμείς την ατάκα μας για ένα εσωτερικό γερμανικό θέμα. Η Γερμανία δεν είναι κανένα διαλυμένο κράτο. Αντιθέτω, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι είναι κράτο δικαίου και οι αρχέ λειτουργούν σύμφωνα με ε, κανόνες αμερόληπτους. Αναρωτιέμαι μήπως αυτό σχετίζεται με την μόνιμη μανία μας για μια κοινή φορολογική πολιτική. Αλλά ίσως είμαι ο μόνος εδώ μέσα που αισθάνεται έτσι. Δεν είναι λίγο περίεργο να ακούμε όλα αυτά τα εξοργισμένα σχόλια περί αποφυγής από ευρωβουλευτές οι οποίοι εξαιρούνται από το να πληρώνουν εθνικούς φόρους εισοδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε το επόμενο ψήφισμα, τον ρόλο της Γερμανικής Υπηρεσίας Πρόνοιας. Τον λόγο έχει ο Μαριάς. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί ο ρόλος της Γερμανικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Παιδιών και Νέων, ο περίφημο Jugendamt, πραγματικά έχει με τη δράση του αυτά τα χρόνια ξεπεράσει τα όρια είναι άπειρες οι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει στην επιτροπή αναφορών. οι γονείς διαμαρτύρονται και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην γερμανία αυτοί οι οποίοι δεν είναι γερμανοί πολίτες και αφορά έλληνες γάλλους κροάτες. έχουμε επανειλημμένα πάρα πολλές καταγγελίες και από τους πολωνούς και υπάρχει μια λογική στο Γιούγκενταμ. εάν ο ένας εκ των γονέων είναι γερμανός πάντοτε να υποστηρίζει αυτή την περίπτωση δηλαδή τους γερμανούς. και αυτό είναι πλέον μια διοικητική πρακτική η οποία εφαρμόζεται χρόνια ολόκληρα. παρεμβαίνει το Γιούγκενταμ μέσα στη λειτουργία του οικογενειακού δικαίου με διακριτικό τρόπο εις βάρος όσων, όσων δεν είναι γερμανοί. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Κύριος σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την γερμανική Jugendamt. Βλέπουμε να υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα συνεννόησης και απόρριψη των υποθέσεων όπου εμπλέκονται αλλοδαπή γονείς, ε, εκεί που οι οικογένειες είναι μικτές. Ε, το Κοινοβούλιο λοιπόν λήφθη του θέματος διότι πάντοτε έχουμε κατά νου τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν πρέπει να σχετίζονται με, με το θρησκεύμα, την ε, καταγωγή, την, ε, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης. Οι πολιτικοί λοιπόν που επιζητούν την εξουσία ζητούν και κάποια προνόμια. Ελπίζω τώρα να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φιλελεύθερο κράτο δικαίου που έχουμε δημιουργήσει δεν μπορεί με την κοινωνική μηχανική που προβλέπεται να καταστρέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί ακριβώς επισημαίνει ένα πρόβλημα αυτό της διακριτικής μεταχείρισης των μη Γερμανών γονέων στην ε, Γερμανία αποτέλεσμα να τους παίρνουν τα παιδιά τους. Αλλά οι πρακτικές αυτές επίσης ισχύουν και σε άλλες ε, χώρες όπως η Ολλανδία. Αυτό παραβιάζει τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έχει επαφή και με τους δύο γονείς εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με τα συμφέροντα του παιδιού. Στην Επιτροπή Αναφορών ε, μας έχουν φέρει αποδείξεις για το ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα παιδιών και γονέων. Παραδείγματο χάρη δεν μπορούν να μιλήσουν την γλώσσα τους. Ε, και έχουμε έναν εκγερμανισμό των ε, παιδιών, ε, κάτι το οποίο μπορεί να καταλήξει στη χειρότερη περίπτωση και σε θάνατο των παιδιών που τα χωρίζουν από τις μητέρες τους. Η Γερμανική Υπηρεσία Πρόνοιας δεν λειτουργεί σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριος Χοκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό. Είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα. Πάρα πολλές ε, αναφορές έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να το δούμε από την σκοπιά του πραγματικού ανθρώπινου δράματος ε, και όχι από τη σκοπιά της πολιτικής ορθότητας. Από ό,τι ακούμε από την Πολωνική Ένωση Γονέων που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό η υπηρεσία αυτή μόνο το 2016 πήρε 77.000 παιδιά από τους γονείς τους δεν ναι, τα βλέπουν επί χρόνια και να τα δουν δεν μπορούν να τους μιλήσουν την ε, γλώσσα τους πριν από λίγα χρόνια μια επιτροπή του Κοινοβουλίου αυτού υιοθέτησε μια επικριτική έκθεση αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή καμία συνέχεια. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή η υπηρεσία αυτή να αρχίσει να λειτουργεί ε, με βάση μόνο το συμφέρον των παιδιών. Σας ευχαριστώ κύριο Σονκέλη, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από την Επιτροπή Αναφορών και είχα εμπλακεί και εγώ στο θέμα αυτό και είχα λάβει κάποιες καλές απαντήσεις ε, στις αναφορές που είπε. Αλλά Δέχομαι βεβαίως πλήρως ότι οι ε, θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους ε, στην γλώσσα τους. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, εγώ και η ομάδα μου καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση γιατί αυτό είναι θέμα κράτους μέλους και είναι υποχρέωση του κράτους μέλους να το επιλύσει. Και Επιτροπή Αναφορών. Επίσης έχει αναφορές και για άλλες τρεις χώρες. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα μαζί χωρίς να εστιάζουμε σε μία μόνο χώρα. Αν και συμφωνώ πλήρως με την αρχή. Σας ευχαριστώ κύριο Σάναν. Ευχαριστώ. Είναι ένα τομέα όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι κάνουμε. Είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, η σχέση μεταξύ ε, γονέων και τέκνων. Είδα ορισμένε καταστάσει στην Επιτροπή Αναφορών και στην ε, εκλογική περιφέρεια που πραγματικά λυπάσαι ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει να συμφωνήσω με το φίλο από το έκτο Σον Κέλλη. Αυτό είναι ακριβώ, επειδή είναι τόσο λεπτό το θέμα, είναι το είδο θέματο που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω των εθνικών δημοκρατικών ε, μηχανισμών και διαδικασιών κάθε χώρα. Για δεύτερη φορά σηκώνομαι για να υπερασπιστώ τη γερμανική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει πω δεν αναγνωρίζω το πρόβλημα. Αλλά ποιοι πρέπει να το επιλύσουν. Αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται πιο άμεσα. Δηλαδή οι αρχέ του κράτου μέλου. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ολοκληρώνονται οι επεξηγήσεις ψήφου για το θέμα αυτό. Και το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Lange Ρουίμπιχ Πόε ε, «Η οδός προς το μέλλον». Η κυρία Κέρτον Ντάλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πολυμερείς κανόνες ε, απειλούνται ε, όπως ποτέ στο παρελθόν. Είναι συλλογική μας ευθύνη να υπερασπιστούμε αυτό το σύστημα, ιδιαίτερα λόγω των επιθέσεων που υφίστανται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εδώ γίνεται πολιτική τη ζούγκλα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε κανένα κράτο μέλο από μόνο του έχουν καμία δυνατότητα να ε, προωθήσουν ένα ε, προοδευτικό μέλλον. Ο ακρογωνιαίος λήθος ε, της πολυμερούς προσέγγισης είναι ο ΠΟΕ. Ο μηχανισμός διευθέτησης διαφορών που έχει είναι ένας από τους λίγους διεθνείς μηχανισμούς που έχει δυνατότητα να επιλύσει διαφορές ειρηνικά. Ξέρουμε ως Ήπειρος στο παρελθόν ότι οι οικονομικές ε, αντιπαραθέσεις πολύ συχνά οδηγούν σε πολιτικές σειράξεις, αλλά ο ΠΟΕ φυσικά δεν είναι καθόλου τέλειος. Πρέπει επιτέλους να αυξηθεί το πεδίο εφαρμογή της δράσης του για να βοηθήσει την ανάπτυξη, τους εργαζόμενους και των περιβάλλον. Για να σώσουμε τον ΠΟΕ πρέπει να τον κάνουμε πιο αποτελεσματικό, να λογοδοτεί καλύτερα και γι' αυτό στήριξα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Ντρογεύσκη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε και στη συζήτηση χθες. Θα θυμάστε ότι το 2008 υπήρξε μια σοβαρή αποτυχία και μάλιστα φιάσκο θα έλεγα όταν εγκρίναμε το πρώτο ψήφισμα που έλεγε ότι ο ΠΟΕ θέλει κάποια μεταρρύθμιση. Για μένα αυτό που είναι ζωτικό είναι ότι στην ε, προηγούμενη δεκαετία ναι ε, έγιναν κάποια πράγματα αλλά ελάχιστα. Στην τελευταία διάσκεψη σε υπουργικό επίπεδο τον περασμένο χρόνο στο Buenos Aires, προέκυψε ότι η διαπραγματευτική λειτουργία του οργανισμού αυτού έχει σταματήσει εντελώ να λειτουργεί. Έχει παραλύσει. Πρέπει λοιπόν να, το σύστημα. να, συγγνώμη, να αλλάξει το σύστημα. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση δεν μπορείτε να πείτε ότι την τελευταία δεκαετία δεν έγινε τίποτα. Όχι. Πολλά όντω έγιναν. Αλλά δεν επαρκούν ούτω ώστε αυτό ο οργανισμό να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ο κύριο Ρόρι Πάμα. Ευχαριστώ. Η εμπορική ιδιοκτησία ε, μειώνεται σε αξία, μειώνεται ε, 25% η λίρα, μειώνεται η τιμή των ε, ακινήτων το ΑΕΠ μειώνεται κατά 8%. Αυτές είναι οι προβλέψεις που γίνονται. Αυτά λένε ότι θα συμβούν στον Ηνωμένο Βασίλειο εάν το Brexit ε, γίνει άτακτα χωρί συμφωνία. ορισμένη εδώ μέσα είναι υπέρ της άτακτης αποχώρησης και ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσουμε μετά με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ, αλλά δεν απαντούν στις πιο προφανείς ερωτήσει αυτοί που τα λένε αυτά. Αν οι κανόνε του ΠΟΕ είναι τόσο τέλειοι γιατί η χώρα μας ε, έκανε τόσο μεγάλη ε, προσπάθεια. Γιατί όλες οι χώρες το κάνουν αυτό για να έχουν συμφωνίες ελευθερου εμπορίου. Όσοι θέλουν ένα σκληρό Brexit ή ένα Brexit χωρίς συμφωνία πρέπει να μας πούνε γιατί θέλουν όλοι οι πολίτες του ΗΠΑ Βασιλείου να γίνουν φτωχότεροι. Όσοι συζητούν για Brexit χωρίς συμφωνία πρέπει να καταγγελθούν. Είναι επικίνδυνες ανοησίες. Ευχαριστώ πολύ. Άλεξ Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή την έκθεση για το πόσο ο ΠΟΕ θα γίνει πιο αποτελεσματικός. Φυσικά οι κανόνες του ΠΟΕ για την πρώτη φορά συζητιούνται στην ε, καθημερινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί αυτοί που είναι υπέρ του σκληρού Brexit μας λένε ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία σημαίνει ότι θα εργαζόμαστε με βάση και θα εμπορευόμεθα με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ. Τι θα σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις που εξάγουν στην Ευρώπη. Θα υπάρξουν δασμοί ενώ τώρα δεν υπάρχουν τεράστια αλλαγή. Θα είχαμε 12% δασμούς για τα ψάρια μας ε, που πιάνουμε στο σάφολ, στο και τα ανταλλακτικά για φορτηγάκια από το Λούτον όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν 10% και 21% για τις ντομάτες μας, το Essex, όταν μπαίνουν στην Ευρώπη. Και θα υπάρχουν και ποσοστώσεις. Θα περιοριστεί και ο όγκος εξαγωγών μας. Και αυτό πριν ήδη αρχίσουμε να ξεκινήσουμε την αδιαπραγμάτευση των 124 ε, εμπορικών συμφωνιών που αυτή τη στιγμή έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κόσμο, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το περήφανο εξαγωγικό μας έθνος θα αποδεκαδιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Μάμικης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΠΟΕ παραμένει ένα υπόδειγμα των εμπορικών κανόνων που γίνονται αντικείμενο διαπραγματεύσει σε πολυμερέ επίπεδο και επιτρέπει στα κράτη που θέλουν να είναι σύγχρονα να δράσουν αναλόγω. Ε, είναι μεταξύ των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση η πολυμερή διαπραγμάτευση ε, και προσέγγιση. Όμω, κάποια κράτη όπω ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε συμπεριφέρονται με τρόπο με αυθαίρετε αποφάσει. Θα πρέπει λοιπόν εμεί να φροντίσουμε το εμπόριο να ε, επιτρέπει ισοτιμή συμμετοχή για όλους. Και Υπάρχουν εδώ εκκλήσει για περισσότερη διαφάνεια στο διεθνέ εμπόριο, ώστε να αυξηθεί η σταθερότητα των εμπορικών ροών. Ε, ιδιαίτερα με απασχολούν για τάξει για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των αρχών του ΠΟΕ, θα πρέπει να αποφύγει την ε, κατάσταση ε, τη εκμετάλλευση των χωρών αυτών, να επιτρέψει στι χώρε αυτέ να αναπτυχθούν ω ισότιμοι εταίροι και να ε, γίνουν από ε, αναπτυσσόμενε χώρε ανεπτυγμένε, όπω εμεί. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε στήριξα το σχέδιο πρόταση των κ. Λάγκια και Ρούμπι για τον εξοχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Καλωσορίζω την έκθεση, γιατί πιστεύω ότι οι αλλαγέ αυτέ είναι ουσιαστική σημασία προκειμένου ο ΠΟΕ να γίνει και πιο ε, σκόπιμο στη δράση του και να προσαρμοστεί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, για να αντιμετωπίσει τι αλλαγέ που απαιτούνται και για τον ίδιο τον οργανισμό. Με αυτό το νομοθετικό ψήφισμα ε, θέλουμε να καλέσουμε να ξεπεραστούν οι δυσκολίε τη Αυτούρκη Συνόδου στον Πένο Άρε τον περασμένο ε, και Δεκέμβριο, μάλλον, και να ληφθούν απόψει για την, τον γύρο διαπραγματεύσεων για τα εμπορικά θέματα. Δεν μπορεί ε, να λαμβάνονται αποφάσει για ε, δασμού στον Χάλιβα μονομερό και να δημιουργούνται εμπορικοί φραγμοί. Θα πρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι παγκόσμιε αξίε των εμπορευμάτων και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να είναι προτεραιότητε που θα λάβουμε υπόψη στην εξέλιξη του ΠΟΕ, όπω είπαμε ο κ. Λάγκια και Ρούμπι. Ευχαριστούμε κ. Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, το θαύμα το μεγαλείο του ελεύθερου Σκεφτείτε την ιστορία του Χόγκογκ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά το 1 τρίτο του Ηνωμένου Βασιλείου το ΑΕΠ του. Τώρα είναι 30% υψηλότερο. Και βάσει τίνο πράγματο, ποιου φυσικού πόρου έχει αυτό το νησάκι. Έχει ανάγκη να εισάγει το πόσιμο νερό του, το ηλεκτρική του ενέργεια και ούτω καθεξής. Όλα τα φέρνει απαλού. Η μαγεία ήταν ότι ήρε τα, τους φραγμούς στο εμπόριο και το έκανε πριν από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μονομερής κατάργηση δασμών και φραγμών. Έτσι μπόρεσε να ανθίσει και να αναπτυχθεί οικονομικά. Ε, έτσι έχει και ένα, ένα από τα υψηλότερα βιωτικά επίπεδα σήμερα σε σχέση με τη δεκαετία του 50. Ε, εκτός του ΠΟΕ και εκτός της Θελωνιακής Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι ανάλογο να βγει πρώτη στην κούρσα των ανεπτυγμένων εθνών στον 21ο αιώνα αυτό που χρειάζεται είναι απλώς ε, να άρουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια και τέλη Ευχαριστούμε ο κύριος Πόλτσακ Ευχαριστώ πρόεδρε Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προαλήσαντα. Υπάρχει εδώ γενικώ συμφωνία. Με την άρση των φραγμών μόνο ωφέλει και το εμπόριο μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτό όμως ε, δυστυχώς δεν λειτουργεί με τόσο αυτόματο τρόπο εάν δεν, υπάρχουν, ε, εάν δεν υπάρχει καλή συνεννόηση μεταξύ των κρατών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτόν τον οργανισμό για το εμπόριο, για να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών του. Εδώ όμως και 10 περίπου χρόνια ο οργανισμός αυτός ε, βρίσκεται σε μαρασμό. Η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, όμως δεν συμμορφούνται με τις αρχές και τους στόχους. Και για να μην μιλήσω καθόλου για το Τραμπ και την κυβέρνησή του, τα βήματα και οι αποφάσεις του, ε, σημαίνουν ουσιαστικά την έναρξη εμπορικού πολέμου. Γι' αυτό υποστήριξα το συγκεκριμένο κείμενό μας, διότι ορίζει κάποιες αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην πορεία μας για το μέλλον του ΠΟΕ. Ευχαριστούμε ο κύριο ε, Μακάλιστα τώρα με την έκθεσή του για τη Σερβία. Το λόγο έχει ο κύριος Σντρογεύσκη για το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η Σερβία ξεκίνησε τις επίσημες διαπραγματεύσεις ε, το 2014 τώρα έχουμε 35 κεφάλαια και 14 έχουν ανοίξει ούτε τα μισά δύο έχουν ε, ολοκληρωθεί μόλις ε, θα ήθελα να τα υπενθυμίσω όλα αυτά για να πω ότι με αυτόν τον ρυθμό η Σερβία θα ταχθεί σε 40 χρόνια η έκθεση θεωρώ είναι πάρα πολύ καλή αλλά όσον αφορά την πρόοδο της ε, Σερβίας για να εφαρμοστούν οι στόχοι ε, δεν είναι ικανοποιητική. Και το χειρότερο το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει πρόοδο στο κράτος δικαίου και την ελευθερία λόγου. Σας ευχαριστώ κύριο Σπόλτσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Σερβία είναι μια περήφανη χώρα με μεγάλη ιστορία και, και η σύγχρονη ιστορία είναι γεμάτη γεγονότα χαοτικά μερικά από αυτά περιλαμβάνουν εγκληματίες ε, και τα λοιπά αλλά νομίζω ότι η Σερβία τα ξεπέρασε όλα αυτά και τώρα βρίσκεται καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δοθούν ελπίδες ε, στις χώρες των Βαλκανίων αλλά άλλες χώρες ε, των Βαλκανίων έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από τη Σερβία οπότε Εάν η Σερβία θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να κάνει ε, περισσότερα βήματα. Σας ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του κυρίου Σόλτες για το κοσφοπέδιο. Τον λόγο έχει ο κύριος Σόσνιατς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Κοσμοπέδιο λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύτιμες συμβουλές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι οι τρομοκράτες πρέπει να επανεντάσσονται στην κοινωνία. Αλλά Λογικό είναι μετά να κάνουν ό,τι θέλουν οι τρομοκράτε γιατί του λέμε άμα σε πιάσουμε, α, θα επανενταχθεί στην κοινωνία, θα το μετανιώσει πικρά. Ε, Κυρίε και κύριοι, ε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επανέλθει η θανατική ποινή. Η ε, επανένταξη κοινωνία είναι ανταμοιβή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κερδίσει κανείς. Και εσεί θέλετε να το δώσετε στους τρομοκράτε. Ο Θεό δηλαδή να φυλάει το κοσφοπέδιο με αυτά που του λέτε. Σας ευχαριστώ. Έκθεση Βάγγελ για την Πουγουδουμού. Κυρία Σόιντροβα, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή γιατί η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην πορεία της προς την Ευρώπη. Είναι από τις πιο προχωρημένες υποψήφιες χώρες, αν και υπάρχουν προβλήματα με την δημοκρατία, με το κράτος δικαίου, για να μην μιλήσουμε για την ε, διαφθορά και τις μειονότητες. Γι' αυτό λαμβάνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει μεταρρυθμίσεις. Θετικό είναι ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Ελλάδα για το θέμα του ονόματος και η έκθεση αυτή λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γκροεύσκη, ε, κατέφυγε στην Ουγγαρία όπου ζήτησε άσυλο. Ελπίζω να εκδοθεί στην χώρα για να φυλακιστεί. Τον λόγο έχει ο κύριος Μαριάς. Τα Σκόπια συνεχίζουν να καπηλεύονται το όνομα της Μακεδονίας μας και της ιστορίας μας ταυτόχρονα ακόμη και με το νέο σύνταγμα το οποίο υιοθέτησαν συνεχίζουν την αλυτρωτική τους πολιτική διότι στο άρθρο 36 συνεχίζουν να αναφέρονται σε δίθεν Μακεδονία και σε δίθεν μακεδονικό λαό. Ταυτόχρονα στο προήμιο του συντάγματος αναφέρονται στην απόφαση της Άσνομ του 1944 όπου εκεί ρητά αναφέρεται ότι υπάρχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του δίθεν μακεδονικού έθνους αυτοδιάθεση του δίθεν μακεδονικού λαού. επομένως παραβιάζεται ακόμη και αυτή η κατάπτυστη συμφωνία των πρεσπών από την πλευρά των σκοπιανών. άρα η συμφωνία των πρεσπών είναι νεκρή και δεν δικαιούται καν η ελληνική κυβέρνηση να τη φέρει και να την καταθέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο είμαι λοιπόν αντίθετος με οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη των σκοπίων στην ευρωπαϊκή ένωση και φυσικά καταψήφισα την συγκεκριμένη έκθεση. ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε το κοινοβουλίο μας ε, επενεί τις ε, προσπάθειες ε, της πουγδομού και της Ελλάδας που κατέληξαν σε μια επίλυση του προβλήματος με το όνομα αλλά η χώρα αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα και όπως και άλλες χώρες στην περιοχή όπως η οργανωμένη τρομοκρατία τα ναρκωτικά, τα όπλα λαθρεμπόριο όπλων κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε επίσης πάρα πολύ χαλαροί σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Στο ψήφισμα λέμε ότι χαιρόμαστε για το ότι ε, συναισθήθη μια διακοινοβουλευτική ομάδα για τα θέματα αυτά. Αυτά τώρα είναι περιτά και τα καταψήφισα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ως μέλος της κοινή ε, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, στηρίζω αυτή την έκθεση. Βεβαίω, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη πριν η Μακεδονία να μπορέσει να ενταχθεί στην Ένωση. Αλλά πρέπει να είναι σαφέ σε οποιονδήποτε θέλει να δει ότι έχει υπάρξει ουσιώδη πρόοδο. Η επίλυση διαφορών, όπω για παράδειγμα το θέμα του ονόματο μεταξύ τη Μακεδονία και τη Ελλάδα, θέλει ε, να υπάρχει πολιτική βούληση από πολιτικού μεθάρου που θέλουν να πούν την αλήθεια στου λαού που επιχειρούν να ε, κυβερνήσουν. Η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά κανένα, ούτε οι εθνικιστέ στη Μακεδονία, ούτε οι εθνικιστέ σε αυτό το σώμα προέτειναν καμία εναλλακτική στη Συμφωνία των Πρεσπών. Απλώς στασιμότητα και αδίέξοδο. Ας ε, χαιρετήσουμε το θάρρος των πολιτικών της χώρας αυτής που ε, ε, χαιρέτησαν αυτή τη συμφωνία και να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος για την ε, δημόσια διοίκηση και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Η Μακεδονία έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας από το 2005 και έχει σημειώσει ουσιώδη πρόοδο έκτοτε. Οι μελλοντικές συνταγματικές αλλαγές με βάση την ψήφο στις 19 Οκτωβρίου είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Οι εθνικιστές δεν προτείνουν καμία άλλη λύση. Πρέπει λοιπόν να επενέσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Τις προσπάθειες που γίνονται για να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ αυτών των δύο κρατών. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα, κάποιο βάρος του παρελθόντος. Πρέπει να γίνουν ε, ε, έρευνες για τα κλίμα του παρελθόντος. Υπάρχει ένα ειδικό συμβούλιο που έχει συσταθεί γι' αυτό και πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει και πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η επόμενη έκθεση που θα συζητήσουμε είναι η έκθεση Φλέκενστάιν για την Αλβανία. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ επανειλημμένα έχω δηλώσει εδώ στο σώμα ότι είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της αλβανίας στην ευρωπαϊκή ένωση. πολύ δε περισσότερο καθώς πλέον συνεχίζεται η καταπίεση της ελληνικής εθνικής μειονότητας της βορείου είχαμε πρόσφατα πριν ένα μήνα τη δολοφονία του κωνσταντίνου κατσίφα από την αλβανική αστυνομία συνεχίζει λοιπόν ε, η αλβανία να αρπάζει τις περιουσίες των ελλήνων να γκρεμίζει τις εκκλησίες να αλλοιώνει τον πληθυσμό στη βόρειο ήπειρο και αυτή τη στιγμή προβαίνει και σε νέα αντίπεινα κόβει το ρεύμα εκφοβίζει όλους τους έλληνες που βρίσκονται στη βόρειο ήπειρο και όλα αυτά για να περάσει το μήνυμα ότι δήθεν θα συνεχίσει αυτή την πολιτική της, την πολιτική της καταπίεσης. Της λέμε λοιπόν ότι αυτά δεν περνάνε και ότι συνεχώς θα την καταγγέλουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι ότου να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου. Γι' αυτό και καταψήφισα την συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος ε, Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Αυτό θα επέτρεπε ένα στενότερο έλεγχο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για, ε, για την εφαρμογή των διαπραγματεύσεων. Εφιστώ την προσοχή σα στην επικίνδυνη τάση ε, αύξησης ε, του, ε, της εμπορίας ε, ανθρωπίνων όντων. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, το αναφέρουμε στο σημείο 18, για να καταστρέψουμε τα δίκτυα των διακινητών, που επίσης διακινούν και όπλα και ναρκωτικά. Στο σημείο 23 μοιάζει να προθείτε με τρόπο ε, ε, που δεν χρειάζεται με αυτές τις αναφορές στα άτομα ΛΟΑΔΙ. Αυτό καταψήφισε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Σελίμοβιτς, παρακαλώ. Η Αλβανία έχει κάνει ουσιώδεις ε, πρόοδους και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το ανταμείψουμε. Γι' αυτό βεβαίω είμαι υπέρ του να κινήσουν ε, ενταξιακέ δραματεύσει του χρόνου. Γνωρίζω βεβαίω ότι έχει γίνει πρόοδο, ιδιαίτερα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, αλλά πρέπει να πούμε ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Ιδιαίτερα εκλογική μεταρρύθμιση, γιατί ανησυχούμε γι' αυτό. Τα θέματα τη διαφθορά, του οργανωμένου εγκλήματο και των σχέσεων καλή γειτονία. Οι μεταρρυθμίσει σε αυτού του τομεί είναι οδυνηρέ, αλλά πρέπει να λάβουν χώρα γιατί είναι ουσιώδει. Το κράτο δικαίου, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση τη διαφθορά πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Με αυτό το στόχο θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε για την, ε, ένταξη, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για να μην υπάρξει πίσω γύρισμα. Ευχαριστώ, ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας αναφέρω ένα σκάνδαλο γιατί ε, μια τροπολογία που δεν ήταν γλωσσική διόρθωση αλλά ε, επέτρεψε να περάσουν σκουπίδια το Πούτιν σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή Ε, είναι λε και έχουμε ε, πραγματικά εμεί ίδιοι επιτρέψει να υπάρχει σκανδαλώδε περιεχόμενο στι τροπολογίε μα. Δεν σηκώθηκαν 40 άτομα για να υποστηρίξουν την αντίρρηση κατά τις τροπολογίες και αυτό ήταν απαράδεκτο και γελίο. Ευχαριστώ. Μαυροβούνιο, έκθεση του κυρίου Τάνοκ, η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θέλω να εξηγήσω γιατί ε, στήριξα την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που έχει ευρωπαϊκές ρίζες όπως οι υπόλοιπε ε, και θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης και είναι ένα κράτο που τα πήγε καλά στι διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στα θέματα τη εσωτερική του πολιτική και αναδιοργάνωση. Τα δικαστήρια έχουν γίνει ανεξάρτη, ε, πιο ανεξάρτητα, η δημόσια δίκηση βελτιώνεται και οι προεδρικέ εκλογέ πήγαν καλά τον Απρίλιο φέτο. Οι πολίτε ήταν ελεύθεροι μπόρεσε να αποφασίσουν χωρί ε, πίεση. Υπάρχουν ακόμα κάποιε ανησυχίε για την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, αλλά παρακολουθούμε στενά τι εξελίξει. Ευχαριστούμε, κύριο Πιετρόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για το ψήφισμα αυτό, την έκθεση αυτή. Ε, και ζήτησα να λάβω το λόγο για το θέμα, διότι υπάρχουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ των εκθέσεων για την ε, Μακεδονία και την ε, Αλβανία και εδώ στο σημείο 22 εκφράζουμε την ε, δυσαρέσκειά μας για την έλλειψη καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Αυτό αναφέρεται σε όλες τις εκθέσεις αυτές, σε αυτή τη σειρά εκθέσεων. Και πάλι στεκόμαστε στο θέμα των παιδιών τα οποία οθούνται στην επαιτία αυτά, ε, τέλο πάντων εντάξει, μπορούν να σημειώνονται, αλλά υπάρχει και άλλη μια ανησυχητική τάση εδώ πέρα. Το κοινοβούλιο μα ανησυχεί πάρα πολύ για τι λεγόμενε μειονότητε. Στο σημείο 34 συγκεκριμένα διαβάζουμε ότι μα ενοχλεί το γεγονό ότι ο σεξουαλικό προσανατολισμό, ε, ο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό δεν γίνεται ανεκτό στο Μαυροβούνιο. Γι' αυτό καταψήφισα αυτή την έκθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λίμοβιτς ε, τώρα έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Τάνεκ. Το Μαυροβούνιο παραμένει στην πρωτοπορία των Δυτικών Βαλκανίων με 31 ανοιχτά κεφάλαια και θα θέλαμε να συνεχίσει αυτή η πορεία. Πρέπει όμως να πούμε ορισμένα πράγματα. Η ελευθερία του τύπου που παραμένει ένα ζήτημα. Οι τελευταίες υποθέσεις δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε χώρα που θέλει να ενταχθεί. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση της ελευθερίας έκφρασης και να καταδικάσουμε τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διακριτική μεταχείριση ΛΟΑΤΚΙ και ΡΟΜΑ και να διασφαλιστεί η διαρευνησή των εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Χάν η ακαδημαϊκή ελευθερία στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον λόγο έχει ε, η κυρία Μάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τις μεταπτυχιακές έρευνες και σπουδές ε, και δεν είναι δυνατόν βεβαίω να μην υπάρχει ποτέ κανένα κίνδυνο. Αλλά πρέπει να δούμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων και των δεύτερων. Πρέπει να επαγρυπνούμε όταν ε, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ανοίγουν παρατήματα σε χώρε που δεν έχουν ελευθερία λόγω. Και τρίτον, πρέπει να δούμε τα του οίκου μα. Στην Ουγγαρία ακυρώνονται τα μαθήματα ε, για σπουδέ φύλου την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα τον καθηγητή Μπέτεκ από το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης. Μου είπε ότι το Πανεπιστήμιο είναι κόμβος ε, και προσελκύει ομιλητές υψηλού επίπεδου, τους οποίους αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία να δουν οι Ούγγροι και θα ήταν πλήγμα η μετακίνησή τους στην Βιέννη. Δεν είναι λοιπόν κάτι το θεωρητικό αυτό. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι θεμελιώδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως θα πρέπει ο πληθυσμός των χωρών με τις οποίες είμαστε σε επαφή να μπορεί να κάνει στι πολιτικές επιλογές και όσο μεγαλύτερη ελευθερία έχουν τα πανεπιστήμια τόσο πιο δημοκρατική θα είναι μια κοινωνία και η δημοκρατική κοινωνία όπως ξέρετε είναι πάντα πιο ειρηνική κοινωνία. Εκτιμώ ιδιαιτέρως ε, τις ε, τροπολογίες των σοσιαλδημοκρατών που ζητάνε η ακαδημαϊκή ελευθερία να είναι μέρος ε, των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Αν υπάρχει περιορισμό στην ακαδημαϊκή έρευνα είναι ένα πρώτο σύμπτωμα ανελευθερίας και θα πρέπει κυβερνήσει να μην παρεμβαίνουν σε σχολεία και πανεπιστήμια και όταν αποτυγχάνει εκπαίδευση, αποτυγχάνουν όλες τις σφαίρες της δημοσίας ζωής και επιπλέον καταλήγει σε μια τεράστια απώλεια οικονομικών ευκαιριών. Οπότε στηρίζω αυτήν την έκθεση και ελπίζω οι διατάξεις της να εφαρμοστούν πλήρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Πάλμερ. Ευχαριστώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο που έφερε την πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Νομίζω ότι η δική μου γενιά μεγάλωσε θεωρώντας ε, δεδομένα κάποια πράγματα, κάποιες ελευθερίες που διασφάλισαν οι προηγούμενες γενιές. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελευθερία των μιμία και ακαδημαϊκή ελευθερία επίσης και στην σημερινή εποχή όπου όλα αυτά τα πράγματα αμφισβητούνται στην εποχή του λαϊκισμού, των ψευδών ειδήσεων Όσοι από εμά πιστεύουμε σε αυτές τις ελευθερίες πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μα Η ακαδημαϊκή ελευθερία έχει μεγάλη σημασία και ο λαϊκισμός και οι ψευδεί ειδήσει, ε, τα ψευδή γεγονότα δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο. Πρέπει να προστατεύσουμε τον χώρο ελεύθερης ακαδημαϊκής έρευνας. Οπότε χαίρομαι για αυτήν την έκθεση, με χαρά την υπερψήφισα και ελπίζω να ακούσουμε τα όσα προτείνει. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο κύριο Σάουρθ. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στηρίζω την εργασία του συναδέλφου μου Καν για αυτή την έκθεση που δυστυχώς είναι αναγκαία. Όσοι έχουμε διδάξει ή έχουμε ε, δράσει ως ερευνητέ στα πανεπιστήμια ξέρουμε ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι πολύ σημαντική. Το κράτος δεν είναι δυνατόν να επαγορεύει τι θα ε, μελετάει ε, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είναι απαράδεκτο και εντελώ ασυμβίβαστο με τι ευρωπαϊκέ αξίε. Θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε σκληρά για να υπερασπιστούμε την ακαδημαϊκή ελευθερία. Αν κάποιο κράτο ή τρίτο κράτο επιχειρεί να την περιορίσει δεν θα, μπορεί δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται ούτε από συνεργατικά προγράμματα ε, του ορίζων Ευρώπη ούτε να χρηματοδοτείται. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατική ελευθερία και από την ακαδημαϊκή ελευθερία και από τις δυνάμεις ε, της αγοράς που για οικονομικούς λόγους απειλούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα μου. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας έγιναν μέσω της έρευνας που δεν είχε καμία προφανή οικονομική ε, ωφέλεια. Πρέπει φυσικά να επερασπιστούμε αυτή τη δυνατότητα καθαρή έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να περάσουμε στην έκθεση για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες. Πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Νίρη Άντα. Ευχαριστώ. Ως γυναίκες ε, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις αλλά σκεφτείτε αν είστε γυναίκα και με αναπηρίες. Ε, είναι πολύ σοβαρότερε οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν. Η έκθεση το εξηγεί πολύ σοβαρά. Υπάρχουν διακρίσει. 18,8 των γυναικών στις, ε, ε, των γυναικών με αναπηρίες ε, προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι άνδρες είναι πολύ περισσότεροι, 35,5%. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τα εργαλεία που ε, περιέχει αυτή η έκθεση. Τα κράτη-μέλη βέβαια πρέπει να τα εφαρμόσουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δίδονται οι σωστές υπηρεσίες στήριξης, να διασφαλίσουμε ισότητα στην εκπαίδευση, την υγεία, τον αθλητισμό. Οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή στην, ε, στις εκλογές για παράδειγμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει επαρκή στήριξη μέχρι στιγμής για να μπορέσουν να το κάνουν. Γι' αυτό καλωσορίζω αυτή την έκθεση Αν μια φορά. Είναι όντω πολύ σημαντικό τα ίδια τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα όργανα αυτά και μάλιστα αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλα τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη-μέλη πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουν την κατάσταση σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να στηρίξω αυτό το ψήφισμα γιατί έχω σοβαρές επιφυλάξεις για ορισμένα τμήματα του κειμένου αυτού ιδιαίτερα τα τμήματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης και ε, παρεμβαίνουν επί των δικαιωμάτων των κρατών μελών είτε για τομείς ε, ηθικής είτε για τομείς ε, υγείας. Προτείνει για παράδειγμα το ψήφισμα να περιληφθεί και ο τομέας της αναπαραγωγικής υγείας Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ε, σημαίνει στην πραγματικότητα να του δίνουμε βοήθεια εκτρώσει. Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη ζωή σε όλε τι μορφέ και των γυναικών και των αγενήτων παιδιών. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε επίση ειδικέ καταστάσει στην υγεία για τα δια, διεμφυλικά άτομα. Δεν είναι δυνατόν. Ε, αυτό το θέμα είναι και αυτό, το θέμα τη αλλαγή φύλου, είναι θέμα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό για τις γυναίκες με αναπηρίες διότι σωστά ε, περιγράφει και μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες ε, το τι γίνεται με αυτό το μεγάλο ρυθμό γυναικών και κοριτσιών 60% όλων των αναπήρων ε, συνολικά και έχουν προβλήματα. Ε, υπάρχει στρατηγική για τους ανθρώπους με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως συνεχίζουν να δυσκολεύονται για την πρόσβασή του στην ιατρική περίθαλψη ή για τα δικαιώματα ελεύθερη κυκλοφορία. Τέτοια προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού ε, είναι Πράγματα που δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια και αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης και είμαι υπέρ του ψηφίσματος, αλλά πραγματικά να θυμίσω ότι το πώς φερόμαστε στους αδυναμότερους, παιδιά και αναπήρους, είναι κάτι που χαρακτηρίζει εμάς τους ίδιους και το κατά πόσο αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας στις κοινωνίες μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα την έκθεση αυτή και θέλω να υποστηρίξω ότι η το πώ ε, δυνατή ηθικά είναι μια κοινωνία φαίνεται από το πώ φέρεται στι αδύναμε ομάδε, τι πιο ευάλωτου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σε συνεργασία με του διεθνεί μα εταίρου να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τη γυναική αναπηρία. Ε, αν δούμε του αριθμού, έχουμε λόγο να είμαστε απογοτευμένοι και να θλιβόμαστε. Είναι 46 εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι, έχουν αναπηρίε, αλλά μόνο 18% ε, μπορούν να, κάνουν, να δουλέψουν ε, ελεύθερα. 44% αντιμετωπίζουν διακρίσει λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Και σε, πολλές, ε, σε πολλού τομεί τη δημόσια και κοινωνική σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πολύ λίγε επιλογέ για τον τρόπο που διαβιούν, για τον είδο ζωή που κάνουν είναι θύματα διακριτική μεταχείριση και φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληρότητα στη μεταχείριση των ανθρώπων αυτών που σχεδόν είναι αποδεκτή. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάμπορσκα. Σα ευχαριστώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα των ε, γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία στην κοινωνία μας είναι ένα πρόβλημα. Η ένταξή τους στην κοινωνία, η κοινωνική τους προστασία είναι στοιχεία που ε, πρέπει να απασχολήσουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες ε, κυρίως έγκυται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία έκπτωση εδώ. Το ψήφισμα μιλάει για την άνευ διακρίσεων πρόσβασή του στο σύστημα κοινωνική ασφάλισης και την αναπαραγωγική υγεία μαζί, δηλαδή πρόσβαση και στις αμβλώσει. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση εδώ σε εθνικό επίπεδο όμως και δεν μπορώ να εγκρίνω το σημείο αυτό. Είναι ε, αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναλογικότητα και η επικουρικότητα και αυτό θα τη σεβόμαστε και εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σόσνιερς τελευταίος αγορητής για σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άλλη μια περίπτωση μια σεξιστική πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν σας καταλαβαίνω. Είστε όλοι τρελοί και δεν βλέπετε. Τι δικαιώματα θέλετε να δώσετε στις ανάπηρες γυναίκες που δεν έχουν οι άντρες, τι θέλετε να πείτε Κάνουμε τώρα ψήφισμα για γυναίκες με αναπηρίες. Τι δηλαδή, θα έχουν διαφορετική πρόσβαση στα κτίρια από ό,τι άνδρες ε, όταν μιλάμε για είσοδο αναπήρων. Σε τι διαφέρουν από τους άνδρες; Στο σημείο επτάλογου χάρη λέγεται ότι οι γυναίκε ε, με αναπηρίες έχουν περισσότερα προβλήματα γιατί ζουν περισσότερο. Μα άμα ζουν περισσότερο από του άντρε ε, που ζουν λιγότερο, ε, πού είναι το πρόβλημά του στους άντρες να επικεντρωθούμε, διότι εκείνοι πεθαίνουν γρηγορότερα. Είναι δυνατόν να τους δώσουμε και άλλα προνόμια. Είναι ήδη προνομίο και αφού ζουν περισσότερα. Είσαστε άρρωστοι. Ευχαριστούμε πολύ. ευχαριστώ πολύ. Ε, Τα πρακτικά των συνεδρίαση θα υπάρξουν στην επόμενη συνεδρίαση. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Εάν δεν έχει κανείς αντίρρηση, θα αποστείλω τι αποφάσεις που λάβαμε στις, ε, στους φορείς όπου πρέπει να απευθυνθούν. Διακόπτη της συνεδρίαση και σα εύχομαι καλό απόγευμα.